Good morning. We can start the meeting. Please, colleagues. Good morning to you all. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, ξεκινάμε τη σημερινή μας συνάντηση. Και προχωράμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε σαν σημαντικότερα σημεία στην μεσια διάταξη τις δύο ψηφοφορίες για μπουζούτιλ γνωμοδότηση και την κάουντις επίσης και τη συζήτηση για την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπές μας για το 2011 με τον κύριο Τσίτσεστερ σαν εισηγήτη και επίση τη γνωμοδέτηση της κυρίας Άουκεν είναι και στο ε, Μποστινάρου και στο κύριο Βάλιαν. Και επίση έχουμε μερικές ε, αναφορές που έχουν σχέση με τις διακρίσεις ε, στη Λιθουανία στη σχολική εκπαίδευση και επίσης προβλήματα σε διάφορες προ... περιοχές και την αναγνωριστική μας, την πούμε έτσι, επίσκεψη στο Βερολίνο και στη Ρουμανία επίσης. Εκεί ζητήθηκε όμως μια αναβολή για την εξέταση στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας. Για τις παρουσίες των αναφερόντων θα είναι παρόντες εκείνοι που έχουν υπογράψει τις ε, σημεία 11, 12 και 13 και αυτό για τη σημερινή πρωινή μας συνάντηση και για την απογευματινή ποιοι θα είναι παρόντες υπογράφοντες των σημείων 16 και 17 και 18. Αυτά λοιπόν. Αν δεν έχουμε κάποια αντίρρηση, τότε ζητάω την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Η μοναδική άλλωστε αλλαγή είναι η αναβολή της συζήτησης για την αποστολή μας στη Ρουμανία. Καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν εγκρίνεται τροποποιημένη με τον τρόπο αυτό η μερίσια διάταξη και ψηφίζουμε και την έγκριση των πρακτικών της συνεδριάσεων στις 27 και 28 Φεβρουαρίου του 2012. Κάποιος κάτι θα ήθελε να πει, κάποια παρέμβαση, κάποια αντίρρηση, όχι. Άρα λοιπόν εγκρίνονται και τα δύο αυτά πρακτικά. Έχουν διανεμηθεί ήδη τα παραρτήματα στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα δε να σας υπενθυμίσω ότι όπως συνηθίζεται εγκρίνονται όπως ακριβώς έχουν διανεμηθεί εάν πριν από το τέλος της συνάντησής μας δεν εκφραστεί μια κάποια αντίρρηση από πλευράς των συναδέλφων. Όχι. Καμία άλλη ανακοίνωση από πλευρά μου και θα ήθελα να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Ξεκινάει η ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε σχετικά με δύο έγγραφα. 20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών και επιχειρήσεων της ενιαίας αγοράς. Ο κύριος Μπουζουτήλ είναι ο εισηγητής μας. Απόνομος. Τώρα, άρα λοιπόν, μια και είναι απόν, ούτε μπορώ να του ζητήσω αν επιθυμεί να λάβει το λόγο. Συνάδελφοι, αν δεν εκφράσετε κάποια αντίρρηση, επειδή είναι απόν ο κύριο Μπουζουτήλ, μήπω θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τη σειρά των σημείων στην ημερήσια διάταξη, να ψηφίσουμε την έκθεση του κυρίου Χιουντή. Λοιπόν, αυτά και περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία του θέματος της έκθεσης του κυρίου Χούντι. Παρακαλώ τον συνάδελφο κύριο Χούντι, μήπως επιθυμεί να λάβει το λόγο, να εκφράσει κάτι πριν να ψηφίσουμε. Δεν είμαι ο κύριος Χουντή, είμαι ο κύριος Τριανταφυλλίδης, Εκπρόσωπο του κύριου Χουντή, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, συμφωνούμε να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Allora. Ξεκινάμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία 1 στην παράγραφο 1. Ταμζάντι. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παραγραφός 1 του κυρίου Χουντή, 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 στην παραγραφό 1 Γιάρ και Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 της παραγραφού 1 πάντα, Μέλτσερ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5, παραγραφός 1, Βαλέζα, σε δύο χωριστά μέρη. Το πρώτο μέρος ψηφίζουμε, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, Κατά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ναι, κατά. Καταπίπτει από τη στιγμή που εγκρίνεται η τροπολογία 1 ή 2. Α, λοιπόν, συγγνώμη, συγγνώμη για την προηγούμενη ψηφοφορία. Το δεύτερο μέρος καταπίπτει. Α, λοιπόν, δεν ψηφίζουμε το δεύτερο μέρος της 5. Τροπολογία 6, παράγραφος 1. Α, ταμπζάντι, σε δύο χωριστά μέρη. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος, υπέρ παρακαλώ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολία 8 στη 2. Χάρτονγκ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται αλλά δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Παρακαλώ, συνάδελφοι, μπορούμε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Τροπολογία 8, παράγραφος 2, Χάρτονγκ υπέρ, κατά, Δεκαοκτώ, τι λέτε. Οκτώ, οκτώ, όχι δεκαοκτώ. Παράγραφος δύο, είπαμε. Τροπολογία 8, παράγραφος 2. Του κύριου Χάρτονγκ είναι η τροπολογία αυτή. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν την ψηφοφορία έχει να κάνει με την τροπολογία 8 της παραγράφου 2 από το συνάδελφο Χάρτογκ. Υπέρ, υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές απορρίπτεται τελικά. Παρα... Τροπολογία 11 στο 2α του κυρίου Χουντή. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική λύση 2 στην παράγραφο 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16, παράγραφος 4. Αλφα, μερκής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 στην παραγραφό 5, μοιράντα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, παράγραφος αλφα του κυρίου Χουντή, με προφορική τροπολογία όμως εδώ Μήπως κάποιος θα ήθελε να προβάλλει αντίρρηση. Όχι, καμία αντίρρηση. Άρα λοιπόν ψηφίζουμε την τροπολογία αυτή, τροποποιημένη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 της παραγράφου 6, Μιράντα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 στην παραγράφου 6 του κ. Χουντή, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 21-7 Χουντί υπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22-7α του κυρίου Χουντί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 παραπας 8 Μιράντα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 παράφος 8 Μέλτσερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 παράφος 9 Χάρτονγκ διαγράφεται το άρθρο αυτό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 παράφος 9 του κύριου Χουντή υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 27. Γιάρκε Αλαβράκου. αφορά πάντα την 9 παράγραφο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 στην 9α του κυρίου Πάξας. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 3 στην παράγραφο 10. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 34 στην παραγραφό 11 Μέλτσερ. Τεχνικής φύσεως υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 35 παράγραφος 9α Γιάρ και Σαλαβράκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 11α Μέρκης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 παράγραφος 12 γιάρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι 38, οι 39 και οι 40 καταπίπτουν 41 τώρα, παράγραφος 12α, τα μπάτζι, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42-13 παράγραφος, γιάρ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 παράγραφος 14, γιάρ, σαλαβράκου, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 Παραφός 14α, πάξας, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45, παραφός 15, μέλτσερ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, παραφός 15, Βέρτμαν, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47, 15α, Μέρκης, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 48 παράγραφος 15α του κύριου Χοντή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τελική ψηφοφορία τώρα σχετικά με την γνωμοδότηση αυτή υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται Ομόφωνη η απόφαση εγκρίνεται ομόφωνα. Ο κύριος Μπουζουτήλ εισήλθε στην αίθουσα Α, για τον κύριο Χουντή. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, η τροπολογία 2 θα έπρεπε να είχε καταπέσει από τη στιγμή που η τροπολογία 3 ενεκρίθη. And therefore amendment number Επομένως καταπίπτει η 2. Okay. Ευχαριστώ πολύ και για την παρατηρήσή σας αλλά και για όλη την εργασία την οποία κάνατε αγαπητέ συνάδελφε. Θα περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία στη, της, επί της επόμενης γνωμοδότησης. Έφτασε και ο συνάδελφος Βουζούτιλ. Και επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησής του. Θέλει να πει δυο λόγια ο κύριος Μπουζούτηλ, όχι. Επομένως ξεκινάμε άμεσα. Ψηφίζουμε την παράγραφο 1 του άρθρου 2, 2 συγγνώμη, πρέντεργαστ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 επί του αρθρού 3 στη πέρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 ε, έχει αποσυρθεί. Συμβιβασμός 1 επί του άρθρου 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 επί του άρθρου 4α Κατά τμήματα ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 επί του αρθρού 5 στη πέρα». Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 επί του 5α χουντί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 9 επί του άρθρου 6 χουντί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 επί του αρθρού 8 Πρέντεργκαστ υπέρ κατά αποχές απερίφη. Τροπολογία 11 επί του 8α ε, Μπέκερ υπέρ κατά η αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 έχει απορριφθεί και επομένως ε, ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδοτήσεως υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή η γνωμοδότηση ομόφωνα. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπουζούτιλ για την ε, εργασία του και επομένως ε, δεν έχουμε πλέον άλλες ψηφοφορίες. Ολοκληρώσαμε το τμήμα αυτό των ψηφοφοριών. Μπορούμε επομένως να περάσουμε στη συζήτηση για, τη, για τα σημεία 7, 8 και 9. Η πρώτη έκθεση είναι αυτή ε, του συναδέλφου Τσίτσεστερ. Πρόκειται δηλαδή για την ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών για το έτος 2011. Κύριε Τσίτσεστερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με χαρά θα σας παρουσιάσω αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης επί των δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας για το έτος 2011. Και θα ήθελα βεβαίως πρώτα απ' όλα να αναφερθώ σε δύο-τρία σημεία του εγγράφου μου, να επιστήσω επ' αυτόν την προσοχή των συναδέλφων και ε, να ζητήσω από τους συναδέλφους να κοιτάξουν και κάποιες από τις πολύ ενδιαφέρουσες στατιστικές της επεξεγηματικής σημείωσης. Um, Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζουμε την απόφαση του, του Κοινοβουλίου ε, σε μια προσπάθεια να αναπτυχθεί στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου μια πύλη που θα αφορά ακριβώς τις, ε, ε, την εργασία μας και τις αναφορές και θα μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των αναφορών. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλουμε να το κάνουμε. Το δεύτερο σημείο αναφέρεται στην παράγραφο 4, όπου επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στην προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών μέσω της επιρροής. Δηλαδή, ε, είναι γεγονός ότι μερικές φορές ε, θα καλούμε τις τοπικές αρχές σε δράση ε, και επομένως να έχουμε την δυνατότητα να προωθούμε τις απόψεις μας αυτές και την πίεση προς τις χώρες. Επίσης υπάρχουν δύο θέματα τα οποία προέκυψαν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του έτους. Πρώτον, οι ανησυχίε οι οποίες αφορούν θέματα ιδιοκτησίας στην Ισπανία. Υπάρχουν αρκετές παράγραφοι που αναφέρονται ε, σε αυτό το ε, ε, ζήτημα. Κυρίως δε η περιοχή της Κώστα είναι, ένα θέμα, είναι μια περιοχή για την οποία πολλές αναφορές έχουν υποβληθεί ε, υπάρχει και το υπενθυμίζω για τους συναδέλφους, ε, υπάρχει για το θέμα αυτό και στην περιοχή αυτή μία διαφωνία ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών όσον αφορά αναδρομική νομική ισχύ ε, κάποιων διατάξεων. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο έχει επανέλθει πολλές φορές. Πέραν αυτού, στην παράγραφο 15, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να διασφαλίσει ότι η οδηγία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα ενισχυθεί. Ε, έχουμε πολλές αναφορές στην Επιτροπή μας σχετικά με, την, ε, με τον αντίκτυπο, δηλαδή με τη μελέτη περιβαλλοντικού αντικτύπου και τον ρόλο που μπορεί να παίξει στη ζωή τους. Αυτές οι εκτιμήσεις βεβαίως πρέπει να συνεχίσουν, αλλά θα πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Αυτά είναι τα σημεία τα οποία θα ήθελα κυρίως να υπογραμμίσω και να επισύρω την προσοχή των μελών ε, σε αυτά. Βεβαίως καλοδεχούμενα είναι τα σχόλιά σας, αλλά θα ήθελα όμως να σας παρακαλέσω να κοιτάξετε με προσοχή και τις στατιστικές που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση, γιατί νομίζω ότι μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τον όγκο της εργασίας που αντίχει αντιμετωπίσει η Επιτροπή Αναφορών την πηγή ας πούμε των αναφορών ε, και τις ανησυχίες ε, των ε, πολιτών που αναφέρονται κυρίως βεβαίως μέσα από τις αναφορές οι οποίες γίνονται αποδεκτές. δίνουμε στατιστικές για την ηθαγένεια των αναφερόντων, για την χώρα ε, η οποία αναφέρεται, την οποία αναφορά η αναφορά δηλαδή. Ε, ε, αναφερόμαστε επίσης σε μια άλλη στατιστική στους θεματικούς τομείς, βασικές αρχές, εσωτερική αγορά, περιβάλλον. Μετά αναλύουμε τις περιβαλλοντικές αναφορές Βλέπουμε αυτές οι οποίες αφορούν ε, τις μελέτες περιβαλλοντικού ε, αντικτύπου ή τα απόβλητα. Ε, επίσης έχουμε αναλύσει μέσω στατιστικών τα θεμελιώδη συγγνώμη, δικαιώματα, είτε είναι προσωπικές υποθέσεις, είτε είναι θεμελιώδη δικαιώματα, δικαιοσύνη, ιδιοκτησία κτλ. Έχουμε επίσης ε, στατιστικές ε, για τις αναφορές ε, σχετικά με την εσωτερική αγορά. Πολύ υλικό υπάρχει και δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλα τα σημεία τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους μας ότι πέρσι 242 ετούντες ήρθαν ενώπιον της Επιτροπής για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν αυτή την δυνατότητα οι αναφέροντες, δηλαδή να μπορούν να έρθουν εδώ και να παραβρίσκονται στη συζήτηση των αναφορών τους. Και ε, για το συνολικό αριθμό των ατόμων που παραβρέθηκαν ε, και τους αναφέροντες δηλαδή που ήρθαν και παραβρέθηκαν στις συζητήσεις και για αυτούς έχουμε συγκεκριμένες στατιστικές αναλυτικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τσίτσεστερ. Ε, νομίζω ότι ο κύριος Βίλαν έχει ζητήσει τον ε, λόγο. Yeah, thank you very much. Και η κυρία Μπασέσκου. Α, η κυρία Όκ. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Τσίστεστερ για αυτήν την εξαίρετη έκθεση. Να υπογραμμίσω μόνο δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, εκτιμώ ιδιαίτερος το ότι αναφέρεστε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων να μην είναι γενικόλογη, αλλά να αναφέρεται σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε απέναντί μας πολίτες ε, και πρέπει να τους αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τότε κανένας δεν θα θεωρήσει ότι είναι σημαντική η δουλειά αυτή τη επιτροπή. Αυτό θα πρέπει να είναι το πρότυπο και για τις μελλοντικές αιτήσιες εκθέσεις. Βεβαίως η εστίαση ε, στα προβλήματα της ε, περιοχής αυτής της Ισπανίας που αναφέρεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και βεβαίως αν έχει υπάρξει παραβίαση της νομοθεσία, θα πρέπει να το ξέρουμε ε, και επίσης ο τρόπος με τον οποίο έχουν αντιμετωπιστεί οι περιπτώσει των ανθρώπων αυτών είναι τόσο καταχρηστικός που σαφέστατα είναι υποχρέωσή μας να βοηθήσουμε, ε, να συμβάλλουμε σε μία ε, διάφανη, ε, σωστή και απρόσκοπτη εφαρμογή του νόμου. Θα πρέπει μάλλον να θεωρήσουμε ότι αυτή, αυτό είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγήν. Γιατί εδώ βεβαίως δεν έχουμε εφαρμογή του νόμου, έχουμε καταχρηστική επιβολή του νόμου. Θυμάμαι ότι πήγα στην ε, ε, Βαλένθια και καθόμουν με τα πόδια μου στη θάλασσα σχεδόν και ε, συζητούσαμε για το θέμα αυτό και ήταν σαφές ότι αυτό το ξενοδοχείο το οποίο είχε χτιστεί στον Αιγιαλό είχε χτιστεί με κατάφορη παραβίαση του νόμου. Και καταλαβαίνω λοιπόν τον μεγάλο ρυθμό αναφορών που λάβαμε για το θέμα αυτό. Αναφέρεστε επίσης ε, και το θέμα των Ρωμά και το θέμα του ECI. Γιατί οπουδήποτε και οποτεδήποτε υπάρχει πρόβλημα διακριτικής μεταχείρισης στην Ευρώπη μας αφορά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει. Ε, please. Ο κύριος Βιλάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Τσίτσεστερ για την υποβολή του κειμένου του και την εισαγωγή του. Όσα ανέφερε σε μεγάλο βαθμό τα υποστηρίζω. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν όπως είπε η κυρία Όκεν, αλλά θα επανέλθει σε ένα σημείο. Θα πρότεινα να προσθέσουμε μία-δύο αιτιολογικές σκέψεις που αφορά τη δική μας ε, εργασία. Γιατί επιτύχαμε κάποιες ε, Βελτιώσει τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει πολύ περιθώριο για επιθυμίες περαιτέρω βελτίωσης. Ένα παράδειγμα. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα δυσανάλογο όταν έρχονται επίγοντα θέματα στην Επιτροπή μας. Να φέρω ένα παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι τον Οκτώβριο του 2013 γίνεται μία αναφορά, θεωρούμε ότι είναι επίγουσα, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε εκεί και μετά μπορεί να μας πει το σώμα ότι μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου του 2014 που είναι οι εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πιστεύω ότι εφόσον είναι κάποια επίγοντα θέματα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μέχρι τις 14 Ιουλίου 2014 να επιφορτιστούν βουλευτές να ασχοληθούν με υποθέσεις ούτω ώστε στις 14 Ιουλίου τη μέρα των εκλογών να μπορούν ε, να αναθέσουν στους διαδόχους της στην Επιτροπή Αναφορών εάν πρόκειται λοιπόν ε, για επίγοντα πράγματα να μην χάσουμε ένα ολόκληρο χρόνο. Δεν είναι δυνατόν επειδή υπάρχουν εκλογές για ένα χρόνο να, να μην μπορούμε να προχωρήσουμε τις υποθέσεις μας. Αυτή η ετήσια έκθεση θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί για να πούμε κάτι σαφές για το πώς περιχαρακώνουμε τη δουλειά μας έναντι των πρωτοβουλειών των πολιτών στην Ένωση και έναντι των Επιτροπών Έρευνας. Έχουμε την έκθεση Μάρτιν αυτή τη στιγμή που ασχολείται με ποια δικαιώματα πρέπει να έχουν ακριβώς οι εξεταστικές επιτροπές. Θα ήθελα επίσης να πούμε κάτι το προσεκτικό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να προκύψουν φθόνοι, αλλά κάτι να πούμε, έστω και επιφυλακτικό, που να λέει ότι για ορισμένες αναφορές θα ήταν καλό να είναι εδώ εκπρόσωπος του κράτους μέλους ή του Συμβουλίου Νομίζω ότι η ετήσια έκθεση ε, είναι ο καλύτερος τρόπος να τονίσουμε αυτό το θέμα. Θέλουμε να έχουμε περισσότερες προφορίες. Όταν έχουμε μια συγκεκριμένη αναφορά, θα πρέπει να θεωρούν ότι εμπλέκονται και οι κυβερνήσεις. Θα πρέπει να μπορούμε να καλέσουμε εκπροσώπους των κυβερνήσεων εδώ, γιατί για πολλές αναφορές ο διάλογος με το Συμβούλιο εφόσον αφορά κάποιο κράτος μέλος η αναφορά είναι η καλύτερη πρακτική. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται για την αιτιολογική έκθεση. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν, να το επιβαρύνουμε με τροπολογίες, αλλά για παράδειγμα στο τμήμα των τίτλων να είναι κάπως ε, αναλυτικότεροι οι τίτλοι σε σχέση με την περσινή και την προπέρσινη ετήσια έκθεση, ούτως ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε ευκολότερα από τους τίτλους περί τίνος πρόκειται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βίλαντα. Η κυρία Βασέσκο έχει το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής μας, όμως να την ευχηθούμε καλά γενέθλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφο Πρέντα, που είναι σκιώδη για αυτή την έκθεση, δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ, ε, γιατί έχει ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Γι' αυτό μου ζήτησε να παρουσιάσω την θέση της ομάδας μας όσον αφορά αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή είναι καλή. Όμως ε, θα θέλαμε να προσθεθεί μια παράγραφος όσον αφορά την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Θα θέλαμε να αναφέρουμε λοιπόν αυτήν την εξωτερική συνεργασία καθώς επίσης και την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με την ε, Κομισιόν ε, και την Πραγματογνωσίνη της Επιτροπής που μας επέτρεψε να έρθουμε σε καλύτερη επαφή και να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα των αναφερόντων. Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε αυτά τα δύο σημεία γιατί εμφανίζονται στις παλιές εκθέσεις εκθέσεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, αναφέρομαι μεγάλη, ε, την μεγάλη αναφορά, την, τον μεγάλο αριθμό συγγνώμη, των αναφορών που αναλύονται τώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μπορούμε να, να πούμε, ας πούμε, ότι ε, βάσει των αλλαγών στις, στους κανονισμούς έχει μειωθεί ο αριθμός των αναφορών ε, πιστεύω ότι ε, το τμήμα αυτό του κειμένου θα πρέπει να αναδιατυπωθεί γιατί δεν είναι αρκετά ισχυρό. Ε, πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει εμείς πρώτοι να αναφέρουμε το θέμα αυτό. Επίσης στο σημείο 4 πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στη συνεργασία με τις εθνικές αρχές καθώς επίσης και τις άλλες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μας βοηθούν στη δραστηριότητά μας. Ε, όσον αφορά τώρα τις ε, ε, ε, αναφορές που αφορούν την Ισπανία. Βεβαίως είναι σημαντικές, αλλά πιστεύω ότι δεν αξίζει τον κόπο σε τόσες πολλές παραγράφους να αναφερόμαστε στα θέματα αυτά. Μία παράγραφος πιστεύω ότι είναι αρκετή. Ε, ο συνάδελφος Πρέντα είχε ανταλλαγή απόψεων και με τον εισηγητή ε, και φρονεί ότι όταν στην αιτιολογική σκέψη λέμε ότι ο ε, μεγάλος αριθμός, ο αυξανόμενος μάλλον αριθμός αναφορών σε σχέση με τα μέσα ενημέρωση σχετίζονται με την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφραση στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία είναι πολύ γιατί είναι υπερβολικό εάν πρέπει να συσχετίσουμε το θέμα με την ελευθεροτυπία, θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε έξι ε, αναφορές για την Ουγγαρία, μία για την Ρουμανία και μία για την ε, ε, Πολωνία, μία για την Γερμανία, μία για τη Σουηδία, καθώς επίσης και μία για την Ιταλία και μία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Επομένως, η ομάδα μου θα ήθελε αυτό το θέμα να το διαγράψει. Εκεί που λέει δηλαδή ότι ο ο αυξανόμενος αριθμός αναφορών ε, που σχετίζονται με τον τύπο μπορεί να εξηγηθεί από τα προβλήματα τα οποία η Ρουμανία και η Ουγγαρία αντιμετώπισαν το 2011. Πιστεύουμε ότι η φράση αυτή ε, δεν ανταποκρίνεται σε πραγματικά περιστατικά και επομένως θα πρέπει να ε, τροποποιηθεί, να αναδιατυπωθεί. Εν πάση περιπτώσει όμως ευχαριστούμε τον κύριο Τσίτσεστερ για αυτήν την ε, έκθεση. Ευχαριστώ. Κύριο Βίλαν, και πάλι έχετε επιθυμεί το... Με συγχωρείτε, κάτι ξέχασα, ο κύριο Βίλαν. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια παράγραφο που να λέμε ότι συνολικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και η χρήση του χρειάζονται περισσότερη παρατήρηση. Ε, θα μπορούσαμε κάθε δύο χρόνια να κάνουμε μια κάποια ακρόαση ή ένα workshop, να καλούμε διάφορα άτομα. Πιστεύω για την Επιτροπή μας είναι σημαντικό να ασχολούμαστε και σε γενικό επίπεδο τα θέματα αυτά. Η κυρία Κενταμέν, δύο μικρά σχόλια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ακρόαση που κάναμε. Ήταν πολύ σημαντική ε, θα μπορούσαμε λοιπόν να αναφερθούμε σε αυτήν την ακρόαση. Και μετά θα είχα ένα σχόλιο για την πρόταση του κυρίου Βίλαντ να συνεχίζουμε την εργασία μας μέχρι τις εκλογές. Αν η Επιτροπή μας δεν έκανε μικροπολιτική ορισμένες φορές, λίγο λιγότερη τουλάχιστον. Νομίζω πως αυτό ήταν καλή ιδέα. Αλλά από ό,τι έχω δει σε ορισμένες χώρες, είναι σαφές ότι η αντίδραση κάποιων βουλευτών εξαρτάται από το εάν πρόσκυνται ή όχι στην κυβέρνηση της χώρας που αφορά η αναφορά. Δεν ξέρω λοιπόν αν με αυτές τις συνθήκες θα τα σκόπιμο να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μέχρι ε, τη μέρα πριν τις εκλογές. Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν θα χρειαζόταν να ξαναδώσω ε, το λόγο στον άλφο Βίλαντ διότι λέει ότι η κυβέρνηση κάθε χώρα παίζει ρόλο στην αντίδραση των βουλευτών. Εμεί είμαστε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκπροσωπούμε ο καθένα αυτού που εκπροσωπούμε και καμιά φορά θα έπρεπε να εκπροσωπούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα που θα πρέπει να συζητήσουμε σε άλλα πλαίσια. Ο κύριο Βίλαντ ε, θέλει να συνεχίσει, θέλει να σχολιάσει αυτά που είπε η κυρία Όκεν, ο κύριο Βίλαντ. Ναι, κατάλαβα σαφώς τι εννοεί άνθρωπο Όκεν και συμμερίζομαι τις επιφυλάξεις της. Η πράσινη είναι, κυρία Όκεν, η πράσινη, κυρία Όκεν, η πράσινη είναι ακόμη σχετικά νεαρό κόμμα. Όταν θα μεγαλώσουν, όταν θα γίνουν ενήλικες, θα συμμετέχουν και αυτοί σε αυτούς τους μηχανισμούς, σοβαρότερα τώρα. Υπάρχουν θέματα που δεν αφορούν τόσο πολύ μικροπολιτικά θέματα Εάν έχουμε αποστολές, για παράδειγμα, για αναζήτηση στοιχείων στην Αυστρία για τη φύση, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο το χειμώνα. Οπότε, εάν δεν μπορέσουμε να το κάνουμε την άνοιξη και το καλοκαίρι πριν τι εκλογέ, περνάει ένα ολόκληρο χρόνο. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε ταχύτατα. Πρόεδρο, ευχαριστώ κύριε Βίλαντ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια από του συναδέλφου, να δώσω το λόγο στην Επιτροπή κύριο Φλόριντ. Ευχαριστώ. Λέει ο εκπρόσωπο τροπεπή. Κοιτάξτε, κύριε Τσίζεστερ, η έκθεση θα μπορούσε να είναι λίγο πιο χαρμόσυνη. Το 2011 τα, πολλά, τα πήγατε πολύ καλά ω Επιτροπή. Ε, Χθε το βράδυ προσπαθούσα να σημειώσω όλα τα επιτεύγματά σα και ήταν υπερβολικά πολλά. Και περιορίστηκα σε τέσσερα. Το πρώτο, αυτό το νέο web interface, πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που αναφέρατε επίσης ήδη, η αύξηση η, στη συχνότητα με την οποία οι αναφερόμενοι έρχονται στην έκθεση και τους συναντάτε, ε, έρχονται στην Επιτροπή και του συναντάτε, αυτό νομίζω ότι είναι πολύ καλό. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Τρίτον, λοιπόν, με την ε, ευφυή χρήση της διαδικασίας προφορική ερώτηση με συζήτηση, η δουλειά σας ε, έχει μπει στις πολιτικές προτεραιότητε του Κοινοβουλίου. Έχετε περάσει πολλέ αναφορέ στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο. Δεν είναι και μικρό πράγμα. Οι αναφερόμενοι να δουν να συζητείτε το θέμα του στην Ολομέλεια και αυξάνει την ε, ορατότητα την έκθεση, της ε, δουλειάς σας και την ε, συνεργασία με άλλες επιτροπές. Και κάτι ακόμη. Στην ημερήσια διάταξη αυτή τη συνεδρία το βλέπουμε συζητάτε συλλογικά, συνολικά δηλαδή, ε, αναφορές που είναι στις βασικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Η καλή διαβίωση των ζώων. Τη στιγμή που η αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή αποστέλει έκθεση στην Ολομέλεια. Άρα είστε στις προτεραιότητες, είστε στην πρώτη γραμμή της ε, δραστηριότητας του Κοινοβουλίου. Θα ασχοληθείτε με το άκτα, με το νερό, την ίδρυυση. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει ε, να μας χαροποιούν. Νομίζω ότι οι εργασίες σας είναι πολύ καλές και θα μπορούσατε να είστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Σας ευχαριστώ. Ή μήπως ο κύριος Τσίσεστερ θα ήθελα το λόγο έτσι για να αντιμετωπίσει και πάλι το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω σε ένα-δυο σχόλια Πρώτα απ' όλα, και να μην το ξεχάσω. Ε, άκουσα με μεγάλη προσήλωση ε, αυτήν την ε, συζήτηση για την ηλικία των κομμάτων. Ε, εγώ προέρχομαι από ένα κόμμα το οποίο θεωρείται ότι είναι το γυρεότερο στον κόσμο. Ίσως αυτό εξηγεί κάποιες από τις απόψεις μας, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα λέει πολλά για την επιβίωσή μας σε αυτόν τον κόσμο που διαρκώς αλλάζει. Από αυτό όμως ξεκινώντας, να πάμε στο ε, ειδικό σημείο το οποίο έθιξε ο Βίλεν σχετικά ε, με την συνέχεια της εργασίας μέχρι τις ε, εκλογές. Βεβαίως εν μέρη είναι σωστό, γιατί αυτό θα ενταχθεί στην χαρά της προεκλογικής διαδικασίας. Ε, αλλά ε, νομίζω ότι συμμερίζομαι και την άποψη της κυρίας Όκεν, δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στη διάρκεια ε, της περίοδου πριν τις εκλογές, γιατί να μην πάρουμε διαφορετικές κατευθύνσεις και προσανατολισμούς και να προσπαθήσουμε με πιο αντικειμενικό τρόπο να δούμε τι σημαίνει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. αλλά όντως μπορεί να διαφανούν κάποιες δυσκολίες ε, όχι τόσο όσον αφορά τις, ε, τη μελέτη των αναφορών, αλλά τις ε, αντιδράσεις κάποιων συμφερόντων που ενδεχομένως μπορούν να μας δημιουργήσουν προβλήματα. Όντως διαφαίνεται εδώ μια δυσκολία. Επίσης, να πω στην κυρία Μπασέσκου, καταλαβαίνω τι λέτε, ε, και ε, μπορούν, μπορεί η άποψή σας να εκφραστεί μέσω κάποιων ε, τροπολογιών, γιατί βεβαίως θέλουμε να βελτιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο αυτή την έκθεση, χωρίς όμως να την κάνουμε πάρα πολύ μακροσκελή. Σχετικά με τα όσα είπε ο φίλος μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο οποίος στην ουσία μου λέει ότι θα πρέπει να είμαστε πιο ευχαριστημένοι για τα θετικά σημεία τα οποία έχουμε ε, αναφέρει. Ναι. Ε, συγχωρέστε με, αλλά ως ε, συντηρητικός εγώ μάλλον τίνω να είμαι πιο προσεκτικός και τα, είμαι πεπισμένος ότι από μόνη της θα λάμψει η αλήθεια όπως και τα θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως μπορούμε να υποβάλουμε κάποια τροπολογία κατά αυτή την έννοια σχετικά και με τη συνεργασία, αν και δεν είμαι ε, σίγουρος ότι πρέπει να το κάνουμε. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να είναι σε θέση να εκμεταλλεύεται κατά κάποιο τρόπο τις δυνατότητες που του δίνει το Κοινοβούλιο. Πάντως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ε, γραμματεία για τη δουλειά, ε, για τη βοήθεια που μου παρήχαν σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης αυτής. Και τώρα να δούμε πώς μπορούμε να ε, βρούμε κάποιο χρονοδιάγραμμα σχετικά με την έκθεση. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Θα σας προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα να σας πούμε ότι μέχρι τις 21 Μαΐου ισχύει η προθεσμία για τις τροπολογίες, έτσι. Τότε λίγη προθεσμία. Εντάξει, συμφωνείτε. και θα ακολουθήσει την κανονική πορεία της αυτή η έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών. Από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλα στοιχεία για το θέμα αυτό, περνάμε στο 8. Είναι γνωμοδότηση για το νόμο περί διοικητική δικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φίλη μου κυρία και να έχει το λόγο. Ναι, θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Ακριβώς για να κρατήσω και ξυπνητούς τους ε, διερμηνείς, τουλάχιστον εκείνους που εργάζονται από τα δανεικά. Εδώ πάνω σε αυτή την ε, έκθεση, μάλλον γνωμοδότηση, να σας πω ότι ιδιαίτερα εμπνευστήκαμε από τις βόρειες χώρες που παίζει σημαντικό ρόλο η διαφάνεια και η ανεξαρτησία των, ε, των κομμάτων και η πολίτες ακριβώς είναι κέντρο των δραστηριοτήτων αυτών και όχι η διοίκηση και ο τρόπος ε, με τον οποίο ενεργεί η διοίκηση είναι ακριβώς ότι προσέχει τον πολίτη της ε, και γίνονται σεβαστοί οι νόμοι, εφαρμόζονται υπέρ των πολιτών. Και τα δύο μέρη, ε, και η διοίκηση και οι πολίτες είναι ισότιμοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δε μια τεράστια πρόκληση. Το 73% των Ευρωπαίων πολιτών υποστηρίζουν ότι τα θεσμικά μας όργανα ε, εκεί παρουσιάζεται διαφθορά. Αυτή είναι η πρόκλησή μας γιατί θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες μας να τρέφουν περισσότερη εμπιστοσύνη στα θεσμικά μας όργανα και να ε, εγγυηθούμε έτσι κάτι το διάφανο το δίκαιο να ισχύσει όπως πρέπει, όπως ακριβώς αναφέρεται και από τη Νέα Χάρτα το άρθρο 41 και 42. Εκεί μια χρηστή διοίκηση θεωρείται σαν ένα δικαίωμα των πολιτών και που το επικυρώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβλέψει τον σεβασμό αυτών των άρθρων της χάρτας της Ευρωπαϊκής. Αυτό αποτελεί δε μέρος της όλης εργασίας μας. Μέχρι σήμερα συζητήσαμε ουσιαστικά αυτά τα soft law όπως τα αποκαλούμε δεν είναι όμως μόνο συστάσεις χωρίς κανένα αντίκτυπο είναι απλά ωραία λόγια φραστικά πυροτεχνήματα που δεν εξυπηρετούν σε τίποτα τελικά χρειαζόμαστε σαφείς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις οι οποίες και να εφαρμόζονται και ακόμα ένα από τα στοιχεία της συζήτησης και με άλλους εισηγητές είναι ότι χρειαζόμαστε σαφείς συγκεκριμένες διαδικασίες για να γνωρίζει κανείς ακριβώς ποιες είναι οι ενέργειές μας και ποια είναι και τα δικαιώματα των πολιτών. Και επίσης θα πρέπει να εγγυηθούμε ακριβώς όταν συζητάμε ας πούμε για διάφορους φορείς ε, που δεν σέβονται αυτά τα δικαιώματα αυτής της ρυθμίσης και δεν είναι αρκετά γοργή στην αντίδρασή τους αυτή η φόρης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισό καλά πρέπει κανείς ε, να βιάζεται, αλλά σημαίνει ότι κάθε διαδικασία σίγουρα θα πρέπει να βαδίζει προς συγκεκριμένους στόχους με μια ορισμένη ταχύτητα. Και θα πρέπει να έχουμε και κριτήρια σαφή, ανεξάρτητα από τις διαφορές ανάμεσα σε πολιτικά κόμματα. Και εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα θέματα όπως ακριβώς ε, η ασφάλεια σχετικά με τα τρόφιμα και διάφορα άλλα που σημειώθηκαν προβλήματα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά χρειάζεται, επαναλαμβάνω για προστή φορά, να είμαστε σαφείς και συγκεκριμένα. Εγώ προσδοκώ μια άριστη συνεργασία για να έχουμε μια θετική έκβαση. Ευχαριστώ κύριε Όκεν, λέει πρόεδρος. Και τώρα το κύριος Γιάννη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά που ήθελα να πει ο Σάντο Μπέγκερ, ο οποίο δεν μπορεί να είναι παρόν. Δύο σημαντικές παρατηρήσεις εκ μέρους της ομάδας μου. θεωρούμε ότι είναι πολύ θετική η έκθεση. Ευχαριστούμε την ε, εισηγήτρια για το συγκεκριμένο κείμενο και γενικά θα υπάρξει συνένεση. Δεν θα υπάρξουν ε, σημαντικά προβλήματα. Στο σημείο 3 μιλάμε για αυτήν την ε, ήπια νομοθεσία, soft law, σίγουρα μόνο με τέτοιου τύπου νομοθεσία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε σωστή διοίκηση. Χρειαζόμαστε και τραχή νόμο, δηλαδή διατάξεις. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο αυτός ο τραχής νόμος πρέπει να συμπληρώνεται από ήπιο νόμο. Αν θέλουμε να υπάρξει νοοτροπία ευγένεια, σωστής διοίκησης, σωστής αντιμετώπισης των πολιτών. Δεν είμαστε όλοι άσχετοι. Ξέρουμε πολύ ε, καλά ότι καμιά φορά ο τόνος κάνει τη μουσική. Το πώς παίζεται ένα όργανο. Δηλαδή ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους πολίτες. Ο πολίτης λοιπόν ε, να θεωρεί ότι είναι καλοδεχούμενος όταν πηγαίνει σε μια υπηρεσία Δηλαδή, να υπάρξουν και ήπιες λοιπόν ρυθμίσεις. Οπωσδήποτε είναι σημαντικές. Και για το 8 αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα. Νομίζω ότι η διαδικασία για πρόσβαση στα, ε, στα κείμενα είναι μία από τις λίγες δεσμευτικές διαδικασίες. Υπάρχει ο κανονισμός 2001 ε, που ήδη από τότε δημιουργούσε αυτή την υποχρέωση για τη διοίκηση. Αλλά ε, θα μπορούσε λιγάκι να μπερδέψει το γεγονός ότι πρέπει αυτή η διαδικασία να προωθηθεί μέσω διοικητικών μέτρων, αφού είναι ήδη νομοθετικά καθορισμένη όταν θα εργαστούμε για τον κανονισμό για την άκτα, επειδή ξέρουμε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις νέες αποφάσεις του δικαστηρίου, Φυσικά δεν πρέπει να ξαναρχίσουμε την εργασία από την αρχή, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στις πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου. Και, και γι' αυτό το σημείο συμφωνούμε με τον εισηγητή. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα. Ευχαριστώ και πάλι την εισηγήτρια. Νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά η έκθεση. Δεν επιθυμεί κάποιος άλλος το λόγο. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μας πει την άποψή του και μετά η εισηγήτρια. Κανείς δεν ζητάει το λόγο. Ε, και πάλι συνάδελφος Σάουκεν. Μία σύντομη απάντηση στον συνάδελφο Βίλεντ. Όχι, στον κύριο Γιάρα, στον Γιάρα. Το πρώτο σας σημείο σχετικά με τον ήπιο νόμο, soft law, είναι αυτό που ακριβώς είχαμε και στην αρχή των υπηρεσιών. Δηλαδή αυτό είναι αρεστό στους πολίτες. Και βεβαίως μπορώ να σας πω ότι εδώ αναφερόμαστε στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα όσα συμβαίνουν στα κράτη-μέλη, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Πρέπει να μας απασχολήσει αλλού και να λυθεί αλλού. Πρέπει να έχουμε σαφές δίκαιο όσον αφορά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, εάν εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να εφαρμόσουμε με τραχή νόμο hard law, strict law, ε, στην ε, πρόσβαση στα έγγραφα ας πούμε, ε, αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί στα δημικά όργανα και τότε ίσως να έχουμε πολλές διαμαρτυρίες των πολιτών. Έχω ακούσει από υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν να λένε ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε την ε, ασφάλεια των μελών της ε, ε, Επιτροπής. Δεν νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αυτό που θα πρέπει είναι να διασφαλίσουμε την καλή συνεργασία με τους πολίτες και την καλή διαβίωση των πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφά Όκεν για το σημείο αυτό και εδώ ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το σημείο 7. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών 2 ε, Μαΐου. Η δε ψηφοφορία έχει προβλεφθεί για τις 19 Μαΐου. Πάμε παρακάτω. Το 9 για τη στρατηγική της ένεσης ε, της νομοθεσίας για την ευμάρεια των ζώων. Ο κύριος Μποστινάρου έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή η γνωμοδότηση αφορά την Επιτροπή Γεωργίας και την ε, καλή μεταχείριση των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων. Προσπάθησα στην έκθεση αυτή να συμπεριλάβω τις ανησυχίες αλλά και τις διαμαρτυρίες των πολιτών έτσι όπως αυτές έχουν εκφραστεί σε πληθώρα αναφορών που μέχρι τώρα η Επιτροπή μας έχει λάβει. Προσπάθησα να αναφέρω πόσο σοβαρό ε, είναι το θέμα, πόσο ευαίσθητο είναι το ζήτημα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή η δημόσια γνώμη στις ε, χώρες μας με μεγάλη προσοχή παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές ή οι εθνικές αρχές αντιμετωπίζουν ε, τα ζώα. Το κύριο πρόβλημα το οποίο προκύπτει από τις περισσότερες αναφορές που έχουμε λάβει, αναφέρει ρητά την ε, έλλειψη σαφούς ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των ζώων. Ε, ε, υπάρχουν επίσης αναφορές ε, οι οποίες αφορούν την κακή μεταχείριση των ζώων, είτε ζώων άγριων είτε ζώων αδέσποτων και κυρίως το θέμα των αδέσποτων στις κεντρικές και ανατολικές χώρες της Ευρώπης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Επίσης, για τα ζώα τα οποία τρέφονται σε αγρικίες, το θέμα της μεταφοράς τους είναι πολύ ευαίσθητο. Αποτελεί αντικείμενο πολλών αναφορών αναφορών, καθώς επίσης και μιας γραπτής δήλωσης ε, που εξέφρασε, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα. Ε, οι πολίτες ε, θέλουν να ξέρουν οποιαδήποτε κατάχρηση σε σχέση με την σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση. Υπάρχουν Επίσης ξέρουμε ότι συνεχίζουν πολλά πειράματα στα ζώα. Όλα αυτά τα σημεία λοιπόν αναφέρονται στην γνωμοδότησή μας η οποία θα σταλεί ε, στην Επιτροπή Γεωργίας. Και βεβαίως η συνεισφορά σας είναι καλοδεχούμενη έτσι ώστε να βελτιωθεί η γνωμοδότηση και έτσι ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται άμεσα για αυτό το ευαίσθητο ζήτημα ευαίσθητο πολύ για την κοινή γνώμη σε όλες τις χώρες αλλά και στη χώρα μου τη Ρουμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο ώρα για την εργασία του, για την εισήγησή του, την έκθεση, την έκθεση αυτή. Τέιλορ. Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Η ευημερία των ζώων, όπως ακούσαμε νωρίτερα, είναι ένα θέμα που είναι στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου, στην Ίντα και στην Τραν. Αυτή τη στιγμή εξετάζεται το θέμα. Η δική μας ανατροπή πρόκειται λοιπόν να υποβάλει γνωμοδότηση. Σωστή αυτή η διαδικασία για να αντικατοπτριστεί το ενδιαφέρον της κοινή γνώμης για το θέμα αυτό. Ως Ευρωβουλευτής της Νότια-Ανατολικής Αγγλίας μπορεί να σας πω ότι αν δεν είναι το πρώτο θέμα που αφορά τις επιστολές που λαμβάνω είναι μεταξύ των τριών πρώτων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ευκαιρία να εξετάσουμε την έκθεση Μποστινάρου και θα μπορούσαμε και να προτείνουμε κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσουμε τη στρατηγική που προτείνει η Κομισιόν για την ευημερία των ζώων και έχω υποβάλει μια σειρά από τροπολογίες. Τώρα δεν θα τις ε, εξετάσω μία-μία, σας χαροποιώ πιστεύω αλλά θα σας πω για τις καλύτερες. Και ελπίζω να συμφωνήσετε και να υπερψηφίσετε σύντομα τις ε, τροπολογίες μου. Η Επιτροπή δεν αναφέρθηκε και δεν διασφαλίζει συνοχή με άλλους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με την ευημερία των ζώων. Για παράδειγμα, το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την βιοπικιλότητα. Χαιρετίζω το στόχο της Επιτροπής να εξετάσει ένα απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο για όλα τα ζώα, όλα τα κατοικίδια και τα ζώα που χρησιμοποιούνται για οικονομική δραστηριότητα. Συμπεριλαμβάνοντας φυσικά και τα κατοικίδια. Τα ζώα συντροφιάς. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί καλύτερα η οδηγία για τους ζωολογικούς κήπους και αν σας ενδιαφέρουν οι ζωολογικοί κήποι υπάρχει μια θαυμάσια έκθεση στο επίπεδο 3 δίπλα στις ταχυδρομικές ε, θηρίδες. Από το Ίδρυμα γεννήθηκα ελεύθερος. Θα ήθελα να υπάρξουν εναλλακτικέ λύσεις στην, ε, στα πειράματα με ζώα και ελάχιστα επίπεδα Καλή διαβίωση για τους σκύλου και τις γάτες και να σταματήσει αμέσως η κοινοτική χρηματοδότηση για τις ταυρομαχίε. Επίσης, καλό να υπάρξουν δεσμευτικές προβλέψεις, να συμπεριλαμβάνεται η καλή διαβίωση των ζώων στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου που συνάπτει η Ένωση με τρίτες χώρε. Και τέλος, καλό, για την συμπερίληψη της βελτίωσης των ε, γαλακτοφόρων, τη, βελτίωση της ευημερία των γαλακτοφόρων αγελάδων και υποστηρίζω την αναφορά που έχει υπογραφεί από πάνω από ένα εκατομμύριο πολίτες που καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για τον περιορισμό της μεταφοράς του χρόνου μεταφοράς ανά ημέρα ζών των ζώων σε 8 ώρες. Με χαρά λοιπόν θα συμμετάσχω στη συζήτηση και ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Τέιλορ, συνάδελφε Τέιλορ, Γιάρ. Ευχαριστώ. Αναμφίβολα, πολύ σημαντικό θέμα. Το βλέπουμε και από τις υπογραφές. Να προσθέσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται πολύ με το θέμα αυτό Ξέρουμε ότι είναι διαμεθοριακό θέμα, δεν σταματάει η προσπάθεια αυτή στα σύνορα. Ως πολιτική δυνατότητα μας δίνει την ευκαιρία να προβάλλουμε νομοθετήματα και μέτρα που να ισχύουν σε όλη την Ένωση. Δεύτερον, αν σκεφτούμε την παγκοσμιοποίηση, δεν έχει έννοια να έχουμε καλή κατάσταση για τα ζώα μας ενώ στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται απέσια πράγματα. Τα 500 εκατομμύρια πολιτών είναι η αναγκαία κρίσιμη μάζα, ούτως ώστε να επιδράσουμε συνολικά στην καλή διαβίωση των ζώων σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι η πρόθεσή μας, αυτή είναι η απέτησή μας και οι πολίτες της Ένωσης αντιλαμβάνονται ότι στρεφόμενοι προς εμάς έχουν επιθυμίες που τις καταλαβαίνουμε Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη δυνατότητα να δράσουμε και νομίζω ότι θα μας υποστηρίξουν και οι άλλες αρμόδιες επιτροπές όπως η Άγκρη. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ε, καμία άλλη παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει το λόγο. Θα ήθελε μήπως κάτι να πει βοηθητικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι. Όχι. Ο στην Μποστινάρου και πάλι μήπως θα ήθελε να κάνει ορισμένες καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απολύτως ημερίζομαι την άποψη του έγκριτου συναδέλφου ε, των έγκριτων μάλλον συναδέλφων ε, και βεβαίως με μεγάλη μου χαρά θα ενσωματώσω στην τελική εκδοχή της γνωμοδότησής μου όλες τις απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα, κυρίως δε για να υπογραμμίσω την απόλυτη ανάγκη όχι μονάχα να υπάρξει νομοθεσία προστασίας των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η άμεση ανάγκη να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε εάν συστηματικά αποτυγχάνουν ε, τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή του ισχύοντος νόμου να ληφθούν, λέω, άμεσα μέτρα έχουμε απέναντί μας ένα ζήτημα το οποίο είναι και λίγο ρουμανικό. Ε, οι πρόσφατες εξελίξεις, ο τρόπος με τον οποίο η κοινή γνώμη αντέδρασε στη χώρα μου με κάνει να είμαι ακόμα πιο ενδιαφερόμενος για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει, ε, ε, ε, λέμε στη Ρουμανία, εάν θες να καταλάβεις το ποιόν του ανθρώπου, δες πώς μεταχειρίζεται τα ζώα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση έτσι ώστε η κρίση για την Ευρωπαϊκή Ένωση να περνάει και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτή μεταχειρίζεται τα ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το σημείο που σίγουρα θα ελκύσει ιδιαίτερη προσοχή και ελπίζω και η Επιτροπή να βοηθήσει ιδιαίτερα στην εργασία του Κοινοβουλίου όπως ο κύριος Τέιλορ υπενθύμησε και να μπορέσει να υποβάλει προτάσεις ή να ευαισθητοποιήσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της προστασίας και της ευμάρειας των ζώων τώρα. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό με τις εκθέσεις, την μέρος αυτό με τις εκθέσεις και πριν να έρθουμε τώρα στις αναφορές ε, για να δούμε στα σημεία 10, 11 αν είναι παρόντες οι αναφέροντες. Διακόπτει ο παρακαθήμενος. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε να ακούσουμε τους αναφέροντες πρώτα. Είναι παρόντες. Καμία απάντηση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και τον λόγο έχει ο πρώτος αναφέρον για τη 16-13 του 2012 2010 από την εταιρεία προστασίας ζών, χλωρίδος και πανίδας Αλάβα Βίκη Μουρ το λόγο έχει... Ποιος έχει το λόγο? Συγγνώμη, συγγνώμη, μισό λεπτό, λέει η Πρόεδρος. Ο κύριος Μάσιμο Πραντέλα είναι τις 825-2011 αναφορές και θα μιλήσει και 16-13 αλλά όλες αυτές οι αναφορές στο θέμα αυτό αφορούν όλες ε, τις ίδιες καταγγελίες για παραβίαση, την αυτή παραβίαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Πραντέλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ λοιπόν, λέει ο κ. Πραντέλα, Μάσιμο Πραντέλα, πρόεδρος της ε, Διεθνούς Οργάνωσης Προστασίας Ζωών η οποία συμπλήρωσε 31 χρόνια ζωής και είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση και συνομοσπονδία εκατοντάδων ενώσεων προστασία ζώων σε όλο τον κόσμο που πρόσκειται στον τομέα πληροφόρησης της, ε, του ΟΗΑ από το 1992. Ο στόχος σύμφωνα με το καταστατικό είναι η προστασία και η αξιοποίηση της φύσης και του περιβάλλοντος και την προστασία των ζώνων απέναντι σε οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Σε 7 Δεκεμβρίου μας πέρασε εγώ για να τονίσω το ότι είναι επίγον να πάρουμε κατεπίγοντα μέτρα για το πρόβλημα αυτό παραδώσαμε μία έκθε, μία αναφορά με 112.683 υπογραφές από Ευρωπαίους πολίτες που ζητούν να μην έχουμε πια στα κέντρα περισυλλογής ζώων, παρόμοια θανάτωση ζώων. Είναι ουσιαστικά ενδιάμεση σταθμή και μετά από δέκα μέρες θανατώνονται. Και ήδη οι δήμοι της Ισπανίας πληρώνουν περίπου 80 ευρώ ανά για να τα θανατώσουν. Είναι πραγματικά ιδιαίτερα αυτό για τους τετράποδους φίλους μας και οι Ισπανοί. Έτσι προσφεύγουν σε αυτήν την θανάτωση. Εκεί ακριβώς, σε αυτά τα κέντρα περισυλλογής για τα δέσποτα σκυλιά αλλά και εργατιά της Ισπανίας. Εκεί υποφέρουν, τα μεταχειρίζονται, τα αγνοεί ο νόμος της Ισπανίας που δεν αναφέρει ρητά το θέμα αυτό των ζώων προστασίας και ε, ε, συντροφιάς αντίθετα με ό,τι συμβαίνει ήδη στην Ιταλία από το 1981 και στα κέντρα αυτά περισυλλογής αυτά παίρνουν κρατικές ενισχύσεις για την ευθανασία στα κατοικίδια ζώα που καμία αρχή δεν ελέγχει με ποιο τρόπο διενεργείται αυτή από κόσμο που υποφελείται ακριβώς πάνω από αυτό προτιμούν να τα θανατώνουν με το πιο σκληρό απάνθρωπο τρόπο και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σκληρές απάνθρωπες αυτές οι μέθοδοι. Τα χτυπούν, τα στραγγαλίζουν, ε, τα θανατώνουν με ασφυξία ε, και δεν υπάρχει κανείς έλεγχος, δεν τα συμπονούν, ε, ναι, σκύλους, γάτες, διακόπτει η πρόεδρος, χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Α, ζήτησε να μην πηγαίνει τόσο γρήγορα ο μιλητής. Και είναι ιδιαίτερα σκληρή και απάνθρωπη η μέθοδος. Επαναλαμβάνω, τα χτυπούν, τα στραγγαλίζουν και δεν ασκείται κανείς έλεγχος, δεν τα συμπονούν αυτά τα ζώα. Πολλές περιπτώσεις σκύλων και γατιών που ενώ ήταν στο θάλαμο αερίων σώθηκαν, δεν πέθαναν επειδή είχαν ε, χώσει τη μουσουδίτσα τους ε, στο τρίχωμα του διπλανού του ζώου και μερικές φορές οι μηθανοί ήδη τα μετέφεραν στα κρεματόρια. Και ένα νευρομικό φάρμακο που προκαλεί παράλυση πολλές φορές χρησιμοποιείται και αργοπεθαίνουν και αυτή η περίπτωση σημειώθηκε στο κέντρο πεσυλλογής του Περτορεάλ. Υποφέρουν τρομερά. Κανείς δεν άντεχε, κανείς δεν αντέχει τα ουρλιαχτά τους με τόσο πόνο και πολλές φορές ε, χωρίς τροφή, χωρίς νερό. Από αυτό πεθαίνουν, είτε από πληγές που δεν τους τις φροντίζουν. Ε, και κάθε μέρα έχουμε και ζώα από ατυχήματα σε αυτά τα κέντρα περισυλλογής, τα οποία όμως δεν τα φροντίζουν. Ε, και μερικές φορές είναι τόσο κακές οι συνθήκες ε, κράτησης φύλαξης που προκαλούν πραγματικά τρομερά προβλήματα στα ζώα. Μετά από την 7η Δεκεμβρίου που μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, οργάνωσή μας έστειλε μία απάντηση και είπε ότι για τον έλεγχο, ο έλεγχος δεν είναι στον τομέα στο οποίο ο οποίος είναι αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί κανείς να αφαιρθεί μόνο στο κείμενο από ό,τι μας έγραψαν. Είναι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη για τα, του 1987 για τα ζώα συντροφιάς. Αλλά δεν τα επικύρωσε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και ένα άρθρο που δεν αποκλείει το ενθανάτωση αυτών των ε, αδέσποτων ζώων μόνο και μόνο για να περιρίσουμε τον αριθμό τους. Επειδή δεν υπάρχει λοιπόν ευρωπαϊκή νομοθεσία η οποία να ρυθμίζει τη διαχείριση όσον αφορά την υγεία και την ευμάρεια των ζώων, αυτό δείχνει ότι είμαστε πολύ πίσω και είναι εντελώς αντίθετο με όσα επιθυμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έχουμε 112.683 υπογραφές διαμαρτυρίες που μέσα σε λίγες εβδομάδες έχουν συλλεχθεί κατά αυτό των κέντρων περισυλλογής αδέσποτων ζώων, αυτά δείχνουν, αποδεικνύουν ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να εχθούν παρόμοια βαρβαρότητα. Γι' αυτό ακριβώς εμείς συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε αυτές οι προθέσεις να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα μέτρα. Χρειάζονται νέες ενέργειες και σε τοπικό επίπεδο για να μπορέσει κανείς να έρθει σε επαφή με τις Αρχές και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις εταιρείες προστασίων ζώων, προστασία ζώων της Ισπανίας. Το επόμενο βήμα για την Διεθνή Οργάνωση Προστασία Ζώων θα είναι ένα δίκτυο συνεργασία με τι τοπικέ ενώσει στην Ισπανία, ώστε να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε μια κοινή πολιτική και να επιτύχουμε τα επιθυμόμενα αποτελέσματα για την ευμάρεια των ζώων. Ποιος είναι ο στόχος μας να αναχαιτήσουμε αυτή την ε, τρομερή κατάσταση και ευχόμαστε όσο γίνεται συντομότερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να υιοθετήσει κάθε νομοθετικό μέτρο για να διακοπεί αυτή η σφαγή και έτσι από τώρα να έχουμε όλες τις αναλύσεις, όλες τις εκτιμήσεις, όλες τις μελέτες οι οποίες θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν με στόχο αυτό το μέτρο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που υποβάλατε την αίτηση αυτή και που την παρουσιάσατε. Λοιπόν, τώρα θα δώσω πρώτα το λόγο σε όλους τους εκπροσώπους των αναφορών, ε, έτσι ώστε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει μία ενιαία παρέμβαση. Ε, γιατί είπαμε ότι το αντικείμενο ε, των, των συγγνώμη, αναφορών είναι κοινό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 σας παρακαλώ, επειδή δεν είναι η μητρική μου γλώσσα, ε, να έχετε κατανόηση. Ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα να μιλήσω. Σας χαιρετίζω, κυρία Πρόεδρε. Ωραία, αρχίζω. Η κυρία Πέντελάιτα είχε κάποιες δυσχέρειες, γι' αυτό ανέλαβα εγώ να την εκπροσωπήσω. Σήμερα αφορά την κατάσταση των ε, αδέσποτων ε, ε, σκύλων στην Ρουμανία. Το πιο εμφανές πρόβλημα, με συγχωρείτε, έχω μία παρουσίαση PowerPoint. το πιο εμφανές πρόβλημα όσον αφορά την κακομεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία είναι η κατάσταση των αδεσπότων σκύλων. Η μαζική θανάτωση των αδεσπότων σκύλων εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται. Χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ε, σκύλων έχουν θανατωθεί έτσι. Τα ζώα ε, πεθαίνουν από πείνα ή σκοτώνονται με παράνομες και ε, βίες μεθόδους. Τα ζώα διατηρούνται σε ε, στρατόπεδα θανάτωσης. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ έχουν ούτως δαπανηθεί. Για παράδειγμα, για παράδειγμα τα δημαρχία δαπανούν 12 1.200 ευρώ για ένα μόνο σκύλο. Συγγνώμη, 200 ευρώ για ένα μόνο σκύλο. Και τη θανάτωση ενός μόνο σκύλου. Κυρίως θανατώνονται για ένα αδέσκοτο σκύλο κατά μέσο όρο δαπανώνται 84 ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι δεν τους δίδεται ούτε ιατρική βοήθεια, ούτε τροφή, δεν έχει σχεδόν κανένα κόστος, με πολύ βάναυσους τρόπους και χωρίς τις νόμιμες ε, τεχνικές θανάτωσης. Ενώ η αντιμετώπιση από μη κυβερνητικέ οργανώσεις και επαγγελματικό τρόπο κοστίζει 20 ευρώ και συνδυάζεται με το ενδεχόμενο υιοθεσία. Και έχουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Μείωση, για παράδειγμα, των αδεσπότων. Παρ' όλα αυτά, η, θανάτωση υγιών σκύλων απαγορεύεται από το 2008. Αλλά παρόλα αυτά χιλιάδες σκύλοι θανατώνονται επισήμως. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί μείωση των αδέσποτων στους δρόμους. Ακόμη και μαζική... Ε, Straight population. Conducted until success... Ακόμη και η μαζική στήρωση δεν έχει ε, δώσει θετικά αποτελέσματα. Η Ρουμανία με βάση την ε, πείρα από την πόλη Ραντία κατάφερε να μειώσει τους σκύλους στην πόλη αυτή από 4.400 και στην πόλη Λουγκάι από 2.500 σε, 2.000, σε 200 μόνο ζώα με μια καλύτερη στρατηγική. Οι ρουμανικές αρχές ασκούν πιέσεις για να συνεχιστεί αυτή η μαζική θανάτωση. Γιατί παρόλο που η στρατηγική αυτή δεν αποδίδει, άρα συνεχίζονται αυτά τα προγράμματα από τα οποία πολλοί κερδίζουν. Αυτή η στρατηγική, λοιπόν, όπως ε, είπα, δίνει τεράστια κέρδη σε διάφορες ε, εταιρείες. Δίδονται λοιπόν πάρα πολλά χρήματα Αλλά το γεγονός ότι τα χρήματα αυτά δεν αποδίδουν σημαίνει πως ε, ε, στην ουσία δίδονται αλλού, αξιοποιούνται για άλλους στόχους. Η εγκατάλειψη βεβαίως και ο βασανισμός και η θανάτωση των ζώων είναι εγκλήματα από το 2008. Αλλά συνήθως ε, ακόμη και όταν γίνονται επίσημες έρευνες δεν αποδίδουν. Παρά το ότι είναι αποτρόπαιη αυτή η βία κατά των ζώων, δεν έχει υπάρξει καμία καταδίκη. Κανείς δεν έχει πληρώσει ούτε καν πρόστιμο. Κανείς δεν έχει φυλακιστεί για σκληρότητα κατά των ζώων. Έχουμε στείλει στην Επιτροπή σας και ε, φωτογραφίες και βίντεο που αποδεικνύουν πώς αντιμετωπίζονται τα ζώα στη Ρουμανία. Η κακομεταχείριση των ζώων όπως και η κακομεταχείριση από τσίρκα και από αγορές γίνεται με την ανοχή των αρχών που έχουν την ευθύνη της προστασίας των ζώων. Στον Ποτουζάνη, για παράδειγμα, σκοτώθηκαν, θανατώθηκαν 230 ζώα το Μάιο του 2011. Ενώ ευθύνη για την ε, διαχείριση των ζώων είναι η ευθύνη του Δημαρχείου σε λίγες ώρες ένας ε, κτηνίατρος θανάτωσε 230 ε, σκυλιά κάτι το οποίο σημαίνει ότι για ε, κάθε θανάτωση χρειάστηκαν 30 δευτερόλεπτα. Έχουμε αποδείξεις ότι δεν υπήρξε σωστή ευθανασία αλλά απλή και κτηνώδης θανάτωση δεν υπήρξε η σωστή σύλληψη των ζώων, η ακινητοποίησή τους και η σωστή χορήγηση θανατηφόρου ενέσεως. Ούτε βεβαίως η χορήγηση αναισθητικού. Για να γίνει σωστά η θανάτωση όμως ενός ζώου χρειάζονται 5,5 λεπτά Οπότε θα χρειαζόντουσαν για τη θανάτωση 230 σκύλων τουλάχιστον 21 ώρες, ενώ δαπανήθηκαν ελάχιστες. Σύμφωνα με τα έγγραφα, μόνο για 31 ε, σκύλους υπήρξε κάποια σωστή διαδικασία. Βεβαίως έχει γίνει ευρέως γνωστή αυτή η θανάτωση 230 σκύλων στον Ποτουζάνη, αλλά παρά το γεγονός αυτό, οι αρχές της πόλης, η αστυνομία, η κτηνιατρική υπεύθυνη και το Δημαρχείο έχουν την ίδια λανθασμένη και ε, στάση άγνοιας. Οποιαδήποτε συζήτηση με τους υπευθύνους αυτούς έχει επιπτώσεις. Δεν μπορούμε πλέον να παρατηρήσουμε, να πάμε να επισκεφθούμε τα κοινοστάσια. Μετά από αυτή τη θανάτωση, όλοι οι νέοι ε, αδέσποτοι σκύλοι, όλοι οι αδέσποτοι σκύλοι που ε, συνελήφθηκαν εκ των υστέρων, έχουν πεθάνει από πείνα, χωρίς καμία δυνατότητα παρέμβασης. Και δεν τους ε, χορηγείται βεβαίως και καμία ιατρική βοήθεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια μη κυβερνητικών οργανώσεων να αποκτήσουν πρόσβαση απορρίπτονται. Οι διάφοροι ψηλά ηθήμενοι ή ψηλά ιστάμενοι στον Ποτουζάνη αρνούνται να μιλήσουν μαζί μας. Ακόμη και διάφοροι που εργάζονται για την κτηνιατρική υπηρεσία στην ε, πόλη αυτή. Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα. Έτσι καταδεικνύεται ε, η λανθασμένη στάση των τοπικών αρχών. Επίσης έχουμε κακομεταχείριση των αγρίων ύπων στο Λίδια. Το Μάιο του 2011 διάφοροι αρμόδια από διάφορους δήμους προσπάθησαν να ε, συλλάβουν διάφορα άγρια ζώα που ζουν στο δέλτα του Δούναβη για να τα δώσουν στα σφαγεία χωρίς να είναι σαφές ε, ποιανού είναι η διοκτησία των ε, ύπων αυτών. Τα άγρια ζώα αυτά συνελήφθησαν με ιδιαίτερα βάναυσες και βίες μεθόδους και τα ε, υποχρέωσαν να μπουν μέσα σε κλειστούς χώρους ε, δέρνοντάς τα. Η μεταφορά τους ήταν παρά, ε, απολύτως παράνομη και παρά τις διαμαρτυρίες που έγιναν στην αστυνομία και τις κτηνιατρικές αρχές δεν έγινε καμία αλλαγή. Μετά από 23 ώρες και παρά το γεγονός ότι ε, ακτιβιστές παρακολουθούσαν τα ζώα μετά από 23 ώρες η αστυνομία σταμάτησε την παράνομη μεταφορά. Όταν άνοιξε η πόρτα του φορτηγού ήταν καταστροφική διαδικασία. Είδαμε για παράδειγμα τα ζώα αυτά να υποφέρουν, ε, να διψάνε τρομερά, να έχουν τρομερές πληγές. Η αρμόδια κτηνατική υπηρεσία της πόλης του ΣΥΑ όχι μόνο αρνήθηκε να στείλει εκπρόσωπο για να διαπιστώσει επιτόπου τι είχε συμβεί, αλλά υπονόμευσε συστηματικά κάθε προσπάθεια διάσωσης των ζώων. Ακόμη και μετά από δύο μέρες, οι αρμόδιοι για την προστασία των ζώων, ακόμη και μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κανένας δεν έχει συλληφθεί για αυτές τις ενέργειες. Κανένας δεν έχει τιμωρηθεί δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση. Η άγνοια και η συνενοχή των αρχών που δεν εφαρμόζουν την αντίστοιχη νομοθεσία είναι κατάφορη. Είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας και για, τα του σκύλους, και για τους αδέσποτους σκύλους. Οι αρχές υγιεινής και εκτινιατρικής λένε ότι θα κάνουν κάτι, αλλά στην πράξη δεν κάνουν τίποτα. Και η κακομεταχείριση των ζώων συνεχίζεται. Ενώ κυρίως ε, προσπαθούν να στραφούν κατά των ε, οργανώσεων προστασίας των ζώων. Να σας δώσω ορισμένα παραδείγματα. Κάποιος που ε, έδιρε μέχρι θανάτου το άλογο του δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα. Άνθρωποι που, ήταν για, άνθρωποι που είναι γνωστοί για πολλά χρόνια για κακομεταχείριση ζώων δεν διώκονται. Κατόπιν βέβαια ορισμένοι από αυτούς σκοτώνουν και ε, ε, άλλους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πολύ. Α, και τώρα και τη δεύτερη παρουσίαση. Είναι γερμανικά η δεύτερη. Θα είναι λίγο καλύτερη.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 εργάζομαι για την οργάνωση ε, γιατροί για τα ζώα αφιλοκερδός. Ευχαριστώ που δίνει δυνατότητα να παρουσιάσω την ε, παρουσίασή μου. Έχουμε μαζέψει 200.000 υπογραφές από όλη την Ευρώπη, κάθε μέρα περισσότερες. Όπου ζητάμε να δημιουργηθεί ένας, ε, να υιοθετηθεί ένας νόμος ε, για την προστασία των ζώων ε, συντροφίας και για τα δέσποτα ζώα γιατί οι εθνικοί νόμοι δεν εφαρμόζονται. Θα γνωρίζετε ότι στη Γερμανία δεν απαγορεύεται η σεξουαλική κατομεταχείριση των ζώων. Αλλά βεβαίω ε, φέρουμε ευθύνη την προστασία των ζώων όπω και των παιδιών. Θα γνωρίζετε ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, τα κυνηγετικά σκυλιά στο τέλο τη ε, περίοδου τα κρεμάνε ούτω ώστε ίσα ίσα να φτάνουν τα πόδια του ε, το έδαφο. Οπότε προσπαθούν να βγουν από αυτό από αυτά τα δεσμά τα σκυλιά ώσπου εξαντλούνται και ε, πνίγονται. Οι κυνηγοί το λένε αυτό ε, παίξιμο πιάνου. Ή αλλιώ ε, του πάνε τα πόδια για να μπορούν να, κυνηγήσουν, να τρέξουν πίσω από του κυνηγού όταν τα εγκαταλείπουν. Στη Ρουμανία τα, δέσποτα, τα δέσποτα τα κυνηγάνε οι μπόγε Για κάθε ζώο πληρώνουν 25 ευρώ. Συνεργάζονται με τα κρεματόρια. Με συγχωρείτε που διακόπτω Μπορεί να έρθει ένας τεχνικός γιατί έχουμε κάποια προβλήματα με την παρουσίαση.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 Στη Ρουμανία τα δέσποτα ζώα, λοιπόν, τα πιάνει ο Μπόγιας και τα σκοτώνει. σκύλο 25 ευρώ, συνεργασία με τα κρεματόρια που τα καίνε, δαπανώνται μέχρι 200. Στην Ιταλία τα δέσποτα ζώα δεν επιτρέπεται να θανατώνονται. Οπότε τα βάζουν ε, σε διάφορα στρατόπεδα χωρίς αρκετή τροφή και νερό, χωρίς ε, κτηνίατρο και για κάθε τέτοιο ζώο πληρώνει το κράτος. Είναι τεράστια επιχείρηση που έχει και συνδέσει με τη μαφία. Σε πολλές χώρες ε, θανατώνονται με αέριο, τα σκοτώνουν ε, με ρόπαλα κτλ. Σας παρακαλώ να δείτε πώς βλέπει ένα παιδί αυτές τις βιαιότητες. Να βλέπει πώς ε, τα χτυπάνε στους δρόμους. Μπορεί να κοιμηθεί καλά ένα παιδί έτσι. Δεν θα χάσει κάθε σεβασμό για τη ζωή. Πώς θα συμπεριφερθεί αργότερα ένα τέτοιο παιδί. Στο ίντερνετ μπορούμε να παρακολουθήσουμε παιδιά να βλέπουν τέτοια πράγματα. Ακόμη και λικόπουλα οι νέες αλεπούδες σκοτώνονται. Έτσι, τα, τους ρίχνουν βενζίνη και τις καίνε. Και βλέπουν παιδιά να παρακολουθούν δεν έχουμε μόνο οικονομική ευθύνη για την κατάσταση. Δεν είμαστε μόνο οικονομική ένωση. Είμαστε και κοινωνική οργάνωση. Πρέπει να είμαστε πρότυπο για πολλέ άλλε χώρε, όχι μόνο στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε τέτοιες αποτρόπες ενέργειες ε, να σταματήσουν. Και διότι τέτοιες ενέργειες ε, επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Σε μια Ευρώπη της διαφώτισης και με προσανατολισμό προς το μέλλον θα πρέπει να υπάρξει ένας νόμος για τα ζώα συντροφίας και τα αδέσποτα. Θα πρέπει να το επεξεργαστούμε σε συνεργασία με τις ΜΚΟ. Βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει νόμος που να απαγορεύει την κακομεταχείριση και τη θανάτωση. Θα πρέπει να απαγορεύονται επίσης οι βασανισμοί. Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι είναι απαράδεκτο να δολοφονούνται και να βασανίζονται τα ζώα. Είναι ευθύνη μα όπως και τα παιδιά τα ζώα. Πολλέ φορές ε, τα μεγαλώνουν και τα εγκαταλείπουν οι άνθρωποι. Και δεν ε, γίνεται, για παράδειγμα, η ενέργειες αυτέ δεν γίνονται κυρίω για λόγου ε, Πρέπει να υπάρξει λοιπόν εναρμόνιση. Ένα παράδειγμα είναι η Βουλγαρία. Όποτε έχουμε αδέσποτα ζώα, όταν για παράδειγμα δαγκώσουν κάποιον, η τοπική πολιτική και άλλοι επίσημοι ζητάνε να επανέλθει ένα νόμο για θανάτωση των ζώων. Ενώ υπάρχει λοιπόν σωστό νόμο για την προστασία των ζώων στη Βουλγαρία, δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά να τίθενται ένα αμφιβόλω οι νόμοι. Διότι δεν μπορούμε να ξαρχίζουμε από την αρχή την εργασία μας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο που να απαγορεύει αυτά τα πράγματα. Η Ευρώπη, είναι, η Ευρώπη είναι πρότυπο για πολλά πράγματα. Γιατί όχι για την προστασία των ζώων. Θα πρέπει να κλείσουν αυτοί οι σταθμοί θανάτωσης. Στο άρθρο 2, δικαίωμα στη ζωή, στη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αναφέρεται ότι κανένας δεν πρέπει να είναι θύμα θανατικής ποινής. Και στο άρθρο 4 λέγεται ότι απαγορεύεται η απάνθρωπη συμπεριφορά και βασανισμοί. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται ταπεινωτικές πίνες. Αυτό πρέπει να ισχύει για όλα τα ζώντα ζώα. Η Ευρώπη είναι ένα τεράστιο ορφανοτροφείο για τα αδέσποτα ζώα. Θέλουμε να υπάρξει προοδευτική Ευρώπη. Δεν είμαστε βάρβαροι. Ζούμε σε ένα πολύ αναπτυγμένο πολιτισμό. Γι' αυτό το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανθρωπιστικό και διαρκή τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να περιοριστεί ε, η μαζική γέννηση τέτοιων ζώων, να υπάρξει ένα σαφές πρόγραμμα στήρωσης, ούτως ώστε να υπάρξει φυσιολογική μείωση των ε, αδέσποτων πληθυσμών. Γι' αυτό κάναμε την αναφορά μας. Θέλουν να υπάρξουν ε, νόμοι για την προστασία των ε, ζώων συντροφίας. Να υπάρξουν υποχρεωτικά προγράμματα ε, εμβολίασης και στήρωσης. Να απαγορευτεί κάθε θανάτωση ζώων χωρίς τις αναγκαίες προϋποθέσεις και να χρησιμοποιούνται ε, μέθοδοι θανάτωσης που να μην προκαλούν πόνο. να υπάρξουν ε, προδιαγραφές για τα άσυλα ζώων, να ελεγχθούν οι προδιαγραφές για τα ζώα κυνηγίου, να απαγορευτεί η κακομεταχείριση των ζώων για ε, πειραματικούς σκοπούς και να εισαχθούν ε, ηλεκτρονικά τσίπ και υποχρέωση εγγραφής των ζώων σε μητρώα. Βλέπετε λοιπόν ότι αν υπάρξει στήρωση των ζώων και ευνουχισμός, μειώνεται ο αριθμός των αδεσπότων. Ακόμη και αν θα κάθε, κάθε έξι μήνες τα αδέσποτα ζώα, ο πληθυσμός διατηρείται. Εάν όμως έχει εισαχθεί ανταυτού πολιτική στήρωσης και ευνοχισμού, τότε έχουμε επιτυχέστερα αποτελέσματα. Αυτή πρέπει να είναι η στάση μας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να υποστηρίξετε την ε, αναφορά μας για να σταματήσουν αυτές οι αποτρόπες ενέργειες μέσω μιας ε, προσπάθειας ευρωπαϊκού νομοθετήματος. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς ε, για τις ε, δύο αναφορές που μας περιγράψατε, καθώς επίσης ε, και τις εικόνες που μας δείξατε. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της, στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χέλεν Κλάιν και μετά στον Τενή Σιμώνη. Παρακαλώ. Madame la Présidente. Κυρία Πρόεδρε, αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να μιλήσω πρώτος γιατί ε, εγώ έχω το θέμα της ε, καλής μεταχείρισης των ζώων στη Γενική Διεύθυνση. Ναι, ναι. Εγώ απλώς είχα καταγεγραμμένα τα δύο ονόματα. Χωρίς μικρόφωνο η Πρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω απρόσμενα. Θα ήθελα όμως να πω καθαρά προσωπικά και σαν κτηνίατρος, γιατί και εγώ και η συνάδελφός μου ε, είμαστε κτηνίατροι, να πω ότι με μεγάλη συμπάθεια ακούω αυτά που ε, αναφέρθηκαν σήμερα εδώ. Ε, πολύ συστηματικά λαμβάνομαι επιστολές για την τύχη, τη μοίρα και την κακομεταχείριση και κακή διαχείριση των αδέσποτων ζώων που θανατώνονται με απάνθρωπους και βάναυσους τρόπους. Όσον αφορά τώρα την αξία ε, και το σοκ το οποίο προκαλούν αυτές οι εικόνες. Να σας πω ότι εγώ κάθε μέρα βλέπω τέτοιες ε, εικόνες, αλλά παρόλα αυτά το σοκ δεν... Ε, το, το, αισθάνομαι το ίδιο σοκ κάθε φορά που τις βλέπω. Η επίσημη λοιπόν απάντηση τώρα. Τι λέει η συνθήκη όσον αφορά την καλή διαβίωση των ζώων. Έχουμε το άρθρο 13 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ρητός αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαιτήσει της καλής διαβίωσης των ζώων όταν διατυπώνουν ή υλοποιούν ενωσιακές πολιτικές ε, και ακολουθεί μια σειρά, ε, ένας κατάλογος των δραστηριοτήτων, εσωτερική αγορά, γεωργία κτλ. Το πρόβλημα είναι ότι τα εγκαταλελειμμένα ζώα δεν ε, αναφέρονται, δεν ε, ε, εμπίπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η συνθήκη λειτουργίας δεν μας δίνει νομική βάση για να παρέμβουμε όσον αφορά την ευζοία των ζώων, την καλή διαχείριση των ζώων. Το άρθρο 13 παραδόξως δεν μας λέει ότι θα πρέπει να κάνει το εξή, το α, το β, το γ, η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλή διαχείριση των ζώων. Λέει απλώς ότι θα πρέπει να διασφαλίσουν την καλή διαβίωση των ζώων βάσει καλών πρακτικών κτλ. Η εγκατάλειψη τώρα των ζώων εμπίπτει καλύπτει στην ε, ενωσιακή πολιτική. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές συζητήσεις με τους νομομαθείς ιδιαίτερος και δεν προκύπτει ε, εξ αρχής ότι υπάρχει τέτοια ε, άμεση επαφή ή σχέση ανάμεσα στη γεωργία ας πούμε και τα εγκαταλελειμμένα ζώα. Πολύ συχνά πρέπει να πω ότι σε πολλές ε, χώρες μέλη το πρόβλημα της διαχείρισης ε, των, ε, των ζώων αυτών αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου, τοπική ή περιφερειακή αρμοδιότητα λοιπόν. Δυστυχώς το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ότι για την ώρα δεν μπορούμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να παρέμβουμε σε θέματα τα οποία δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακρηγορώ, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε πολλά επιχειρήματα τα οποία αφορούν επιχειρηματολογία των αναφερομένων, καθώ επίση και των επιστολών που δεχόμαστε εμεί. Γίνεται λόγο ε, στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την προστασία ε, των Ζών συντροφιά, Pet, ε, Pet Convention. Πρόκειται για μια συνθήκη η οποία έχει προετοιμαστεί από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Στο παρελθόν ασχολήθηκε το Συμβούλιο τη Ευρώπη με την προστασία των Ζών και υπάρχει ειδική διάταξη για την προστασία των ζώων συντροφιά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συνθήκη δεν έχει ενσωματωθεί στο Ευρωενουσιακό δίκαιο δεν έχει κυρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως ε, υπάρχουν χώρες οι οποίες την έχουν κυρώσει, αλλά άλλες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν την έχουν κυρώσει. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε για αυτούς που έχουν κυρώσει την συνθήκη αυτή, ε, δεν ε, αφορά αρμοδιότητα ή υποχρέωση μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγξει την ορθή εφαρμογή αυτής της συνθήκη. Και οποτεδήποτε και αν και εφόσον έχει κυρωθεί. Α πούμε, η Ισπανία δεν την έχει επικυρώσει. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των διεθνών της ε, δραστηριοτήτων εργάζεται, συνεργάζεται και με την ε, Παγκόσμια Οργάνωση της ε, Υγείας των Ζώων. Είναι η ΟΗΕ η οποία εργάζεται και για θέματα προστασίας των ζώων και επομένως έχει εκπονήσει μία σειρά καλών κατευθυντηρίων γραμμών. Κυρίως μία κατευθυντήρια γραμμή που αφορά τη διαχείριση των... Euh, τον των αδέσποτων ε, ζώων, την οποία έχουν ενστερνιστεί πολλές ε, οργανώσεις προστασίας των ζώων και η ΟΗΕ ίδια βεβαίως και την οποία εμείς ε, εντόνω στηρίξαμε. Εκεί ε, προβλέπεται ε, μια συγκεκριμένη πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο να μπορεί κανείς να πιάσει τα ζώα αυτά, να τα διαχειριστεί, να τα στηρώσει, να τα ευνοχήσει και με την δυνατότητα θανάτωσής τους, εάν και εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο, αλλά με μεθόδους οι οποίες είναι αποδεκτές και οι οποίες δεν είναι βάναυσες. Για μία ακόμα φορά λέω ότι Όλα τα κράτη-μέλη γνωρίζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, γιατί είναι όλες οι χώρε μας μέλη της ΟΗΕ, ε, αλλά ε, δικιά τους αρμοδιότητα είναι η υλοποίηση αυτών των αρχών. Ε, σε περιφερειακό επίπεδο η ΟΗΕ προσπαθεί να προωθήσει τις δραστηριότητε της, αλλά εμείς απλώς μπορούμε να στηρίξουμε την ΟΗΕ σε αυτές τι διεργασίε τη και διαδικασίε και αυτό κάνουμε άλλωστε. Τέλος, να πω ότι το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2010 ε, ε, ε, είχε ήδη διατυπώσει ε, προτάσεις, συστάσεις ε, για την ευζοία των ε, σκύλων και των γατών κυρίως. Επίσης, υπό Βελγική Προεδρία υπήρξαν κάποιες προτάσεις σχετικά με τα αδέσποτα ζώα. Το σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών έτσι ώστε να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενωσιακό επίπεδο με τα αδέσποτα ζώα. Απλώς κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση που θα αφορά τελικά την κύρια ευθύνη που έχουν οι ιδιοκτήτες ε, και ε, ε, υπάρχει ας πούμε μία σειρά συνοδευτικών μέτρων π.χ. ένα ιστότοπος που λέγεται Carrot Dog και που δίνει προτάσεις σχετικά με την καλύτερη διαχείριση των ζώων. Τώρα και βάσει των συμπερασμάτων του 2012 θα υπάρξει και μία νέα ε, οδηγία όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση, τη μεταχείριση μάλλον των ζώων συντροφιά, τα οποία ε, προσφέρονται στο εμπόριο. Εδώ θα γίνει λοιπόν μία μελέτη, αξιολόγηση αντικτύπου, για να δούμε εάν μπορεί κάτι να γίνει και για τα δέσποτα ζώα. Δυστυχώς όμως είμαι μάλλον απεσιόδοξος, διότι τα δέσποτα ζώα ε, δεν αποτελούν αντικείμενο ε, συναλλαγής και μάλιστα ε, δεν υπάρχει καν δυνατότητα ένταξής τους στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες. Αυτό δυστυχώς είναι το μήνυμα που μπορώ να σας στείλω. Δεν είναι πολύ θετικό. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο μας δίνει τα χέρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ουσιαστικά επιβεβαιώσατε τα όσα ήδη είχε συμπεριλάβει σε επιστολή επιτροπή πέρα από την εισαγωγή με ορισμένα προσωπικά στοιχεία τα οποία και εγώ εκτιμώ. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι, ξεκινάει η συζήτησή μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολυάριθμες αναφορές αποτελούν σαφή ένδειξη ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πραγματικά ανησυχούν για το πώς αντιμετωπίζουμε σκυλιά στην Ευρώπη και όπως ακριβώς από αρκετούς ε, ε, εισηγητές υπόθηκε είμαι κατά και εγώ κατά είμαι κατά τη σκληρότητα τη απάνθρωπη μεταχείρισης. Και εδώ έχουμε τις περιπτώσεις των κέντρων περισυλλογή ε, αδεσποτών ζώων στην Ισπανία και στη Ρουμανία όμως και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και ειδικότερα στη Νότια Ευρώπη. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει μια ρύθμιση νομοθετική σχετικά με αυτό και γι' αυτό ακριβώς τα κράτη-μέλη έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για το τι κάνουν με αυτά τα αδέσποτα ζώα για να δουν ποια είναι αυτά τα αδέσποτα και ενδεχόμενα να τα θανατώνουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κύρωσε την Ευρωπαϊκή Χάρτα, την Ευρωπαϊκή Απόφαση για την Προστασία των Ζώων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η σύμβαση αυτή δεν απέκλειε τη θανάτωση, πάντως ε, η κύρωσή της θα αποτελούσε ένα θετικό βήμα για αρκετά κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ορισμένε ρυθμίσεις για τα ζώα, αλλά αυτό έχει να κάνει με την διατροφή τους ε, για τα ζώα στους ζωολογικούς ε, ανθρώπους για τα εργαστήρια, για τη μεταφορά τους, για την σφαγή τους, για τα βοηδή, για τις ε, οτόκους όρνηθες, για τα αγριαπτηνά, για τα ζώα. Και δεν υπάρχει όμως μια πραγματική ρύθμιση που να αφορά τον καλύτερο φίλο του ανθρώπου που είναι ο σκύλος. Είναι 100 εκατομμύρια τα ζώα συντροφιάς σκυλιά και γατιά που ζουν ε, σε ευρωπαϊκά σπίτια με ευρωπαίους πολίτες. Ε, οι Ευρωπαίοι όμως δεν διαθέτουν μια σχετική ρύθμιση για τα ζώα που είναι περισσότερο σε επαφή μαζί τους. Και σε μια αναρώτημά μου για την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ουκρανία, παρόλο που δεν είναι κρατός ανέφερε και σε αυτό η Επιτροπή. Ε, είπε στην απάντησή της, όπως υπενθύμησε ακριβώς πριν από λίγο η Επιτροπή, ότι δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στα αδέσποτα ζώα και στο περιεχόμενο του άρθρου 13 της Συνθήκης της Σαβώνας που λαμβάνει έτσι υπόψη της τα ζώα. Εδώ, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό το 26 της 2011 ε, αναφορά, ζητήσαμε από την Επιτροπή την παρέμβασή της ε, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει ανάγκη για μια ρύθμιση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διάθεση για κάτι παρόμοιο. Θα πρέπει να δειχτεί αυτό σε μια εργασία ακριβώ στην ημερήσια διάταξη που είναι στρατηγική για την ευζοία των ζώων 2012-2015 για την περίοδο αυτό. Οι γνωμοδοτήσεις κλπ. είναι στην Γεωργική Επιτροπή, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και σε πολλές άλλες επιτροπές περιλαμβάνεται προς εξέταση το θέμα αυτό είναι σημαντικότατο για μας τους συμβολευτές για να δείξουμε ότι η πολιτική βούληση για μια ρύθμιση για αυτά τα ζώα συντροφιάς θα πρέπει τα σχετικά μέτρα να προβλεθούν στα πλαίσια αυτής της γενικής ε, σημαντικής στρατηγικής. Μια ρύθμιση που κατά τη γνώμη μου και των Ευρωπαίων πολιτών τον δείχνουν καθαρά και αναφορές θα πρέπει να υπάρχουν ρυθμίσεις για την εκτροφή των ζωών, προγράμματα στήρωσης, Εμβολιασμό με μικροτσίπ να υπάρχει μια αναγνώριση των ζώων και μια απαγόρευση της θανάτωσής τους. Είναι σημαντικό αυτό η ρύθμιση, αλλά δεν είναι το παν. Θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τα κράτη-μέλη γιατί δυστυχώς και τώρα σε πάρα πολλές ρυθμίσεις, παρόλες τις ρυθμίσεις, αυτές δεν εφαρμόζονται, δεν γίνονται σεβαστές όπως θα έπρεπε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζανόνε. Ο κ. Μποστινάρου τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνουμε να συγκρατήσει κανείς τη συγκίνησή, τη συγκίνησή του ε, όταν βλέπει εικόνες σαν αυτές που μόλις είδαμε. Ε, πραγματικά αισθανόμαστε ταπείνωση ε, όταν βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Είναι σαν να βλέπουμε εικόνες από τον Ταχάου ή από την Σρεμπρενίτσα είναι, πρόκειται για εικόνες σφαγής, για εικόνες ε, άκρατης της ε, βίας. Μα σοκάρουν λοιπόν αυτές ε, οι εικόνες και εμένα με σοκάρουν προσωπικά. Και εγώ έχω, τι να σας πω, είμαι φιλόζωος, έχω ένα ροτβάιλερ, έχω τρεις γάτες, αγαπάω πάρα πολύ τα ζώα. Και μπροστά σε τέτοιες βαναυσότητες πραγματικά σοκάρομαι και εξανίσταμε. Ε, και ε, ε, βάσει μιας ευτυχού συγκυρίας εγώ είχα υποβάλει ήδη μια έκθεση την οποία παρουσίασα σήμερα για το θέμα αυτό. Οπωσδήποτε η κατάσταση είναι επίγουσα και χρήζει παρέμβασης. Αλλά για μένα είναι εξαιρετικά επώδυνο γιατί είμαι Ρουμάνος βουλευτής και η χώρα μου έχει σταθεί στο ειδόλιο του κατηγορουμένου επανειλημμένα για το θέμα αυτό. Εγώ ε, θέλω να στηρίξω μια ενωσιακή πολιτική, αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα γιατί δεν την παρέχει η συνθήκη λειτουργίας τη Ευρωπαϊκή Ένωσης και ότι δεν ε, επιβάλλει ε, η συνθήκη οποιαδήποτε υποχρεωτική κίνηση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Επομένω, παραμένει αδρανής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι, ε, κυρία Πρόεδρε, επισκεφθήκαμε το Βουκουρέστι το Νοέμβριο και πήγαμε και στην Επιτροπή, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο Υπουργός και η ομάδα του αναφέρθηκε σε δύο αναφορές σχετικά με την κακή μεταχείριση των ύπων στο Δέλτα του, Δήμου, του, Δι, του Δούναβη συγγνώμη, ε, καθώς επίσης και την κακομεταχείριση των αδέσποτων σκυλιών. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά στην ουσία ήταν σαν να γελιοποιήθηκε το ζήτημα αυτό. Ένας ε, από τους ομιλητές, ας πούμε, τους συνομιλητές μας ε, είπε ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν το δικαίωμα ε, ζωής και ότι και τα ζώα έχουν το ίδιο δικαίωμα επίσης η Ρουμανία βεβαίως θα πρέπει να αναφερθεί σε αυτές τις δύο αναφορές τις οποίες ακούσαμε σήμερα. Πρόκειται για μία χώρα η οποία συστηματικά δεν ε, εφαρμόζει την καλή ε, μεταχείριση των ζώων. Και μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος στην ε, Δημαρχία του Βουκουρεστίου έχει ένα πρόγραμμα για το Βουκουρέστι ε, το οποίο δεν είναι και ιδιαίτερα καλό. Το κύριο σημείο του μάλιστα είναι ότι θα ξεφορτωθεί όλα τα αδέσποτα σκυλιά στο Βουκουρέστι. Δεν αναφέρεται όμως ο τρόπος και δεν αναφέρεται και το ζήτημα της καλής μεταχείρισης των ζώων σε αυτή την προσπάθεια εξάλληψης ας πούμε των ε, των αδέσποτων ε, ζώων στο Βουκουρέστι. Καλή την πίστη βεβαίως, εμείς μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα κάνει μια καλή ε, κίνηση, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ε, και από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ε, θέλουν την, ε, την λιτότητα είναι αυτοί οι οποίοι τελικά θα δημιουργήσουν προβλήματα στον κόσμο. Ξέρουμε αυτή η λιτότητα που οδηγεί. Οδηγεί σε μείωση των φαρμάκων, οδηγεί σε μια ελλειπή πολιτική η οποία μάλιστα θα εφαρμοστεί τυφλά και δεν θα λάβει υπόψη την προστασία των ζώων. Προστασία των ζώων η οποία οποία εν παρόδο μπορούμε να πούμε ότι είναι ανύπαρκτη στην Ρουμανία και γι' αυτό καταλήγουμε σε αυτές τις μαζικές δολοφονίες των ζώων. Πρέπει να το βροντοφωνάξουμε και να το φωνάξουμε και προς αυτούς ε, οι οποίοι θέλουν να στηρίξουν την, ε, ε, να στηρίξουν την λιτότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει οι αναφορές αυτές να παραμείνουν ανοιχτές. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να τις αναφέρουμε ε, και στην, ε, στη, στην, στην επιτόπου επίσκεψη, διερευνητική επίσκεψη που κάναμε. Επίσης, επειδή είδαμε αυτές τις τρομερές φωτογραφίες, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και σαφή απάντηση από τις ρουμανικές αρχές ζητώντας κυρώσεις. Ευχαριστώ πολύ να υπενθυμίσω την προηγούμενη συζήτησή μας όπου μιλήσαμε για το πόσο επίκαιρο είναι το θέμα αυτό της προστασίας των ζώων. τρει παρατηρήσεις. Η ευθύνη των ανθρώπων για τη φύση, για τα ζώντα όντα είναι σαφής. Υπάρχει λευκή βίβλος διότι ο άνθρωπος έχει φτιάξει το περιβάλλον όπως είναι τώρα. Έχει διαμορφώσει το περιβάλλον. Είναι η ευθύνη μας για όλα τα ζώα και φυσικά και για τα ζώα συντροφίας. Καταλαβαίνω επίσης ότι είναι απόλυτα σωστό από πλευράς θεωρητικής ότι το θέμα αντιμετώπισης των ζώων θα μπορούσε ε, να είναι αρμοδιότητα κάθε περιοχής. Γιατί ίσως να αντιμετωπίζεται από τις Βρυξέλλες, να είναι υπερβολικά συγκεντρωτικό. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν λειτουργεί αυτή η κατάσταση. Βεβαίω, συμφωνώ με την θεωρητική αντιμετώπιση τα κράτη-μέλη να ασχοληθούν. Αλλά στην πράξη δεν λειτουργεί. Όταν ήμουν ε, εθνικός βουλευτής είχαν επισκεφθεί τη Ρουμανία πριν την ένταξή της. Το θέμα δεν ήταν ε, η νομοθεσία. Η Ρουμανία έχει ένα από τα καλύτερα νόμο προστασία ζώων στην Ένωση. Το θέμα είναι η εφαρμογή του. Τίθεται λοιπόν αυτό το θέμα. Δεν μπορούν ή δεν θέλουν ή δεν έχουν επαρκείς πιστώσεις για να αναλάβουν ορισμένα μέτρα, όπως για παράδειγμα ευνοχισμού. Αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο όμως, αυξάνεται το πρόβλημα, αυξάνονται οι διαστάσεις του, οπότε σιγά σιγά τα δέσποτα ζώα είναι κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τότε αρχίζει η θανάτωση, που δεν θα χρειαζόταν. Δεν θα ήταν αναγκαία η μαζική θανάτωση, αν είχε υπάρξει μία σωστή αντιμετώπιση, αν είχε περιοριστεί η αναπαραγωγική δυνατότητα των ζώων. Υπάρχουν δυνατότητε. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν. Ρωτάω λοιπόν την Κομισιόν πώς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Τα κράτη-μέλη αντιστέκονται. Δεν θέλουν ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτά που γίνονται δεν είναι δυνατόν να γίνονται σε ένα πολιτισμένο κράτος. Παρ' όλα αυτά αρνούνται, αντιδρούν. Όχι, δικό μας θέμα, μην αναμειγνύεστε. Ρωτάω λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήταν το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε να πούμε ότι αν πρέπει να θανατωθούν να θανατωθούν με το σωστό τρόπο. Ανώδυνο τρόπο. Δεν θα μπορούσε η Κομισιόν να επηρεάσει. Δηλαδή να πει κάθε χώρα, ας το κάνει όπως θέλει, αλλά όχι με μεσαιωνικό τρόπο, χωρίς να θέλω να θίξω το μεσαίωνα. Νομίζω ότι τότε αντιμετώπιζαν καλύτερα τα ζώα. Είναι αναξιοπρεπές αυτό που συμβαίνει. Απαράδεκτο. Γι' αυτό θα ευχαριστούσα τον συνάδελφο Μποστινάρου να διατηρήσει την Επιτροπή όπως λέει. Πρέπει ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να αναλάβει η Ένωση πρωτοβουλίες και να έχουμε αρμοδιότητες ούτω ώστε να πούμε εντάξει να ορίζεται τις λεπτομέρειες όσον αφορά τη σύλληψη και θανάτωση αλλά να είναι σωστός τρόπος για τα ζώα τα οποία είναι χρήσιμα σε εμά, υπάρχουν προδιαγραφές. Αλλά για τα δέσποτα ζώα δεν ισχύει τίποτα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως, αν δεν υπάρχει σωστή αντιμετώπιση της αναπαροϊκής δυνατότητα των ζώων, δεν πρόκειται ποτέ να λύσουμε το πρόβλημα. Η κατάσταση αρμοδιοτήτων, λέω στην Κομισιόν, είναι ιδιαίτερα λυπηρή να μην είναι ανοιχτό το θέμα, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε στην Ευρώπη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στα κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα κακά νέα. Τα καλά νέα τώρα είναι ότι η κοινή γνώμη, οι πολίτες δεν αποδέχονται όλο και περισσότερο την κατάσταση και θέλουν αλλαγή. Ευχαριστούμε τον κύριο Γέρο Imaginile cu aceste animale și filmele Αγαπητέ Άλφε Μποστινάρου, συμφωνώ απόλυτα. Οι εικόνε που είδαμε είναι αποτρόπες και αυτέ που είδαμε στι 24 Μαρτίου ήταν επίση απαράδεκτες σκοτώθηκε ένα παιδί στη Σουτσάβα από ένα δέσποτο σκύλο κοντά σε ένα νεκροταφείο, ενώ γύριζε σπίτι από το σχολείο. Βεβαίως, τα ζώα έχουν δικαίωμα στη ζωή, αλλά και οι άνθρωποι. Αγαπώ τα ζώα, έχω πάρει σπίτι μου δύο αδέσποτα ζώα και να με καταλάβετε. Τα αδέσποτα αυτά ζώα, επειδή δεν υπάρχει λύση για αυτά, στην Ρουμανία σκοτώνουν ή τραυματίζουν άτομα και αυτά περνάνε στον τύπο και αν σας είχαμε δείξει εικόνες από παιδιά που τα έχουν σκοτώσει ή ακροτηριάσει ή παραμορφώσει ε, αδέσποτα ζώα ε, θα είχατε την ίδια αντίδραση. Οι αρχές της Ρουμανία από όλες τις ε, πολιτικές τάσεις και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση κάνουν ό,τι μπορούν για να εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται σωστά, όπως είπε και ο κύριος Γιάρ. Και προσθέτω ότι διατηρώ τη γνώμη μου. Το πρόβλημα αυτό είναι εθνική αρμοδιότητα, όχι κοινοτική. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μιράντα έχει το λόγο. Η συνάδελφος Μιράντα, πρόεδρε ευχαριστώ με τις πολιτικές αποφάσεις και με την εφαρμογή των ρυθμίσεων. Έχουμε και το δολογικό κανόνα, την ηθική αυτών των αποφάσεων. Πέρα από το δεν υπάρχουν αρμοδιότητες, θα πρέπει να ληφθούν σε μια πιο προχωρημένη κοινωνία, όπως είπε ο κύριος Γιάριο, ο κύριος Μποστινάρου στην προηγούμενη ακριβώς έκθεση. Δεν υπάρχει ένας δεοντολογικός κώδικας ε, για παρόμοιες εγκαταστάσεις ε, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, ακριβώς και από την τοπική διοίκηση που δεν υπάρχουν και πόροι και μερικές φορές και σε εγκαταστάσεις όπου δεν ασκείται κανείς έλεγχος και ούτε και αρμοδιότητες για εκεί. Λοιπόν, ε, αμέλεια από πολλά κράτη-μέλη. Θα ήθελα να προτείνω κάτι, μια και υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που αυτή την ε, ε, ΠΕΤ δεν την έχουν υιοθετήσει. Μήπως εδώ θα μπορούσαμε να στείλουμε μια επιστολή, έτσι, ενημερωτική επιστολή, ζητώντας από τα κράτη-μέλη που αυτή τη σύμβαση δεν την υιοθέτησαν, την υιοθετήσουν. Επίσης και θα αποτελούσε και μια πολιτική χειρονομία στην κατεύθυνση αυτής της ηθικής και αυτής, αυτού του δεοντολογικού κώδικα. Και από τη Γαλλική από που προέρχομαι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις σημαντικές. Ε, αυτά τα δέσποτα ζώα, τι γίνεται θα μπορούσε να αποτελέσει και μια αναλλακτική λύση σε αυτή τη δυνατότητα. Παλαβαίνουμε και πολλές ενώσει ακριβώς οι οποίες προστατεύουν παρόμοια υιοθέτηση ζώων και ακόμα από πλευρά ομάδα μας θα έπρεπε να διατηρήσουμε ανοιχτέ αυτές τις αναφορές. Αυτό ζητάω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ αγαπητή συνάδελφε Μιράντα. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι η Επιτροπή έχει το λόγο για μια απάντηση. Και στο τέλος οι αναφέροντες. Η εκπρόσωπος... Μισό λεπτό να δούμε. η Έλεν Κλάιν, η οποία δεν είχε λάβει προηγουμένω το λόγο αυτό, από ό,τι καταλάβει δεν επιθυμούσε να λάβει το λόγο. Μήπω τώρα ναι. Παρακαλώ, μήπως θα μπορούσατε τώρα να λάβετε το λόγο. Ναι, σε όλους καλημέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ενδεχόμενα θα ήθελα να λάβω το λόγο για να εξετάσω το σημείο 10 της ημερησίας διάταξης μια αναφορά που έχει σχέση και με το πρόβλημα του ελέγχου του πληθυσμού των ζώων ε, για σκυλιά και γατιά και ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα αυτά ε, αδέσποτη σκύλη στην Ισπανία ας πούμε ότι ε, ότι την χάνουν ε, παράνομης εξαγωγής. Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι οι Ισπανικές αρχές δεν είναι υιοθετούν ε, δεν σέβονται την νομοθεσία ακριβώς την ευρωπαϊκή για αυτά τα ζώα, τα δέσποτα και το εξετάσαμε αυτό το θέμα, δεν θα ήθελα να επεκταθώ αλλά παρακαλώ μία παρένθεση να κάνω. Δεν άκουσα καθόλου τι γίνεται με τον έλεγχο αυτού του πληθυσμού μέσω μιας διαχείρισης και των πτωμάτων τους. Τι γίνεται αν υπάρχουν, μάλλον όχι, τα, τα, τα, σκουπίδια. Τι γίνεται, γιατί αυξάνεται αυτός ο πληθυσμός σαν Επειδή υπάρχουν σκουπίδια, άρα λοιπόν ένας ευνοχισμός ή μια αυτανασία, εντάξει, καλό το μέτρο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει από κοινού να καταφέρουμε να ελέγξουμε αυτά τα σκουπίδια που υπάρχουν στα κρατημέλη και στα οποία τρέφονται αυτά τα δεσποτα ζώα. Αυτά λοιπόν. Και επίση λένε αναφέροντα ότι ακριβώς δεν εφαρμόζουν την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εξαγωγή αυτών των ζωών, των αδέσποτων και ότι θεωρείται σαν παράνομη. Αυτό το εξαγωγή σημαίνει μια κάποια διακίνηση πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας προς ένα άλλο κρατος μέλος. Εμείς διαθέτουμε σχετική νομοθεσία ευρωπαϊκή που καλύπτει παρόμοια κίνηση, κυρίως για ζώα όπως ε, τα σκυλιά και τα γατιά που σε αυτή την περίπτωση θεωρούνται σαν ζώα ε, συντροφιάς και είναι μη εμπορική διακίνηση στη μια περίπτωση που έχουν να κάνουν με την 8 του 2003 ε, συμφωνία Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και τι προβλέπει όταν τα ζώα συντροφιάς ακριβώς συνοδεύουν τους κατόχους τους οι οποίοι μετακινούνται, ταξιδεύουν και δεν προορίζονται ούτε για πώληση ούτε για αλλαγή ιδιοκτήτη, τότε θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε απαιτήσει αυτού του κανονισμού και ακούσατε βέβαια ότι οι σκυλοί θα πρέπει να έχουν μια ταυτότητα, να τύχουν εμβολιασμού και τα γατιά βέβαια και οι πληροφορίε αυτέ θα πρέπει να δίδονται σε αυτό το α το πούμε διαβατήριο του ζώου συντροφιά. λοιπόν σε περίπτωση μη κλασική εμπορική συναλλαγή, Ακριβώ συνοδεύουμε αυτά τα ζώα τον κάτοχο τα μετακινείται τώρα από τη στιγμή που έχουμε μια μετακίνηση κυβέρνηση που δεν ισχύει αυτό, τότε έχουμε μια εμπορική συναλλαγή και έχουμε ανακείμενο το 92 65 ε, του, του 85 που λέει που προβλέπει παρανασχάρη ότι χρειάζεται μια εξέταση κλινική 24 ε, ώρες πριν από την αναχώρηση να δούμε ακριβώς ποια πορεία εμπορική ακολουθείται στο κράτος μέλος προορισμού. Και η ανακοίνωση αυτή γίνεται με ένα πληροφορικό σύστημα, το TRAS, το ίχνος. Εδώ λοιπόν ε, στις εμπορικές αυτές ε, μετακινήσεις ε, λαμβάνονται υπόψη αυτή η έλεγχη και πριν από την εξαγωγή και πριν την άφηξη στον προορισμό και μάλιστα γίνονται κατά, χωρίς διάκριση και επίσης υπάρχουν δυνατότητες επιβολής κυρώσεων ε, σε σχέση ακριβώς με τις παραβιάσεις που γίνονται και που θα ανακαλυφθούν ενδεχόμενα σχετικά με αυτές τις μετακινήσεις και για τις αναφορές αυτές ε, θα πρέπει βέβαια κανείς να καταφέρει να αποδείξει και να προσδιορίσει τι ακριβώς, πώς μετακινείται το ζώο, με τι στόχο στα πλαίσια της εξαγωγής, της παράνομης όπως αποκαλείται ε, σκυλιών και γατιών αδέσποτων και επίσης η ανάλυση αυτή γίνεται μόνο σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γιατί από τη στιγμή που η κυριότης του ζώου αποδεικνύεται στο διαβατήριο αυτό πριν από τη μετακίνησή του Πρόκειται για μία ας πούμε εμπορική μετακίνηση. Κάπως μπερδεμένα ίσως σας φαίνονται αυτά. Αλλά δεν μπορούμε έτσι τόσο εύκολα να κρίνουμε για τι περίπτωση πρόκειται ότι είναι πραγματικά παράνομη αυτή τη μετακίνηση του ζώου. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και δεν μπορούμε να ασκήσουμε έτσι γενική κριτική πάνω σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Ακριβώς ε, για να απαντήσω στο δεύτερο μέρος, ε, όσον αφορά την προστασία ζώων για τα δέσποτα ζώα, προσπαθούμε να το σκεφτούμε και ανέφερα προηγουμένως ιδιαίτερα σε μια περιφερειακή επιτροπή της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων ε, και βέβαια ορισμένοι επικεφαλής κτηνίατροι που ανησυχούν για αυτή την κατάσταση και θα ήθελαν λεπτομερέστερη εξέταση. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν με, διεθνή οργάνωση οργάνωση μπορούμε να συνεργαστούμε για να δούμε ακριβώ τι μπορούμε να κάνουμε για τα δέσποτα ζώα. Συγγνώμη βέβαια, φτάσαμε έγκαιρα, αλλά εσείς προχωρήσατε λίγο γρηγορότερο σε αυτή τη στρατηγική. Σχετικά με τη στρατηγική, τι θα προτείνουμε, στη... κάτι το νέο νομικά και θα προσπαθήσουμε εκεί να δούμε πώς αυτά τα ζώα συντροφιά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν, βέβαια ανάλογα με τις συνθήκες με διάφορους όρους και θα υποβάλουμε μια νομική πρόταση το 2014 και ακριβώς για λεπτομερέστερη εξέταση θα το δούμε αυτό αν τα ζώα συντροφιά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε, ένα γενικότερο, σε μια γενικότερη δημησία αλλά εκφράζω επιφυλάξει ιδιαίτερα στα αδέσποτα ζώα γιατί είναι τοπικής αρμοδιότητας περισσότερο. Έτσι. Αλλά θα προσπαθήσουμε πάντως εμείς μιας ευρύτερης πολιτικής έτσι, ε, πληροφόρηση κλπ. Όπως το είπαν και οι βουλευτές και οι αναφέροντες εδώ οι σχέσεις με τα ζώα είναι μια αντίληψη των σχέσεων που έχουμε με τους διπλανούς μας και στα πλαίσια αυτό αποτελεί μέρος δε μιας ε, ενός συλλογισμού για τις σχέσεις μας επαναλαμβάνω γενικά. Βέβαια Υπάρχουν ε, μέσα εργαλεία, ας τα πούμε έτσι, αντιμετώπισης, θα μπορούσαν να μας ωφελήσουν πάντως για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε γενικά τα ζώα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και στο σημείο αυτό τώρα ε, δίνουμε το λόγο για δύο λεπτά για τον καθένα, για όσους υπέγραψαν ε, τις αναφορές. Ο κ. Πραντέλα. καταρχάς. Ναι, ευχαριστώ να πω μερικά πράγματα συντροματικά σε περιπτώσεις ε, ατόμων που σε επιτίθενται ζώα και τους ακροτηριάζουν πολλές φορές. Εγώ είμαι από το Μιλάνο και μια γέλια δέσποτων σκύλων σκότωσε ένα ηλικιωμένο άτομο. Το πρόβλημα δεν είναι τα σκυλιά. Είμαστε εμείς και οι αρχές που δεν μπόρεσαν να λύσουν το πρόβλημα των αδέσποτων σκυλιών. Δεν φταίνε ούτε οι άνθρωποι ούτε τα σκυλιά. Συλλαμβάνονται τα ζώα. Ε, και ακριβώ επειδή υπάρχουν διάφορε ενώσει και πιέζουν, υπάρχει ένα νόμο που το απαγορεύει στην Ιταλία, δεν θανατώνονται. Αυτοί τα σκυλιά, τα αδέσποτα που ζούσαν σε αγέλη ακριβώ ε, ε, ενώ συνελήφθησαν στην αρχή, μετά δόθηκαν ε, σε ορισμένους και εδώ υπάρχουν και ενώσεις προστασία ζώων, αλλά είναι βέβαια και εκπροσπεύουν το ενδιαφέρον εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που απαιτούν ή επιθυμούν μια νομοθεσία που να εγγυάται την ευζοία των ζώων και τον σεβασμό που οφείλουμε στα ζώα, όπως επίσης και για τα σκουπίδια των ατάλων. Εάν λυθεί το πρόβλημα της σωστής διαχείρισης των ζώων αυτών, θα υπάρξει μια λύση. Δεν υπάρχει άλλο σύστημα, κάτι ακόμα. 2014 ακούω, 2015 το ένα το άλλο. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Μέχρι το 2014 θα έχουμε και πολλά άλλα ζώα που θα βρουν το θάνατο και θα υπάρξει και ο κίνδυνος για αρκετούς ανθρώπους στους οποίους θα επιτεθούν ζώα και που θα βρουν το θάνατο αυτό. αυτούς. Γι' αυτό χρειάζεται όσο γίνεται συντομότερα μία αλλαγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. θα ήθελα να επανέλθω στα όσα μας είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Έχει δίκιο. Όταν λοιπόν ε, ε, εμείς εκφράσαμε τον προβληματισμό μας, μας είπαν ότι δεν υπάρχει ενωσιακή αρμοδιότητα. Ε, και μας είπαν ότι δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αίτημα των κρατών μελών. Θα πρέπει τα ε, κράτη-μέλη να δηλώσουν ότι ανικανότητα αντιμετώπιση του προβλήματος και μετά να επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω δεν θα σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ζώα, να δημιουργήσει όμως ένα πλαίσιο που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Εάν υπάρξει ένας τέτοιος νόμος, τότε έχει δικαίωμα να παρέμβει η Ένωση. Δεν θέλουμε δηλαδή να σωθούν τα ζώα, απλώ να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για να μπορεί να παρέμβει η Ένωση. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω, ίσω να μην πέρασε. Φυσικά στις χώρες μέλη υπάρχουν, μέλη υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν τηρούνται. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά θα έπρεπε να τηρούνται οι νόμοι και στα κράτη-μέλη, που αποτελείται από κράτη-μέλη. Το... Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο το Βατικανό και τα χανσιατικά κράτη. Τα κράτη-μέλη αποτελούν την Ένωση. Το κόστος αναφέρθηκε επίσης. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, αναφέρθηκε. Ο ευνοχισμός είναι φθηνότερος από την ε, θανάτωση. Τουλάχιστον με βάση αυτά που δηλώνονται ως κόστος ε, θανάτωσης. Βέβαια η αλήθεια είναι αλλιώ. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική η θανάτωση όπως ο ευνουχισμός. Γιατί τότε τα ζώα δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Τρίτο σημείο τα παιδιά που τους επιτίθενται, που τους επιτίθενται αδέσποτα ζώα. Φρικόδες αυτό. Αλλά το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο ότι θα ανατώνονται φρικοδός, αλλά προηγουμένως κακομεταχειρίζονται. Τους πετάνε πέτρες, ακόμη και παιδιά, τους χτυπάνε, τους σκύλους αυτούς με ρόπαλα. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο γίνονται επιθετικοί σκύλοι. Κάποιοι μπορεί να είναι επιθετικοί από τη φύση τους, αλλά ορισμένες φορές απλώς αμήνονται και τότε λέγεται κτηνώδη συμπεριφορά τους. Δεν ισχύει αυτό. Τα θέματα που αναφέρθηκαν, η επιρροή που έχει αυτή η καθημερινή θανάτωση ζώων στους δρόμους, στα παιδιά, η επίδραση στην ε, συμπεριφορά τους, στην ψυχική τους διαμόρφωση, είναι τρομερό θέμα. Πολύ σημαντικό. Διότι με αυτόν τον τρόπο το λέω κάπως ε, υπερβολικά, αλλά δημιουργούμε βίαιους ανθρώπους. Θα μπορούσε να αποδειχθεί και επιστημονικά αυτό. Πολλοί που κάνουν εγκλήματα, που δολοφονούν ε, ανθρώπους, που δολοφονούν πολλούς ανθρώπους, είναι γνωστό ότι ξεκίνησαν κακομεταχειριζόμενοι ζώα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο. Να το έχετε υπόψη σας. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Οι αναφορές βεβαίως παραμένουν ανοιχτές. Νομίζω ότι είναι ομόφωνο το αίτημα αυτό. Φρονώ πως η Επιτροπή ε, Αναφορών ε, έχει οπωσδήποτε μια, αυτή την πολιτική εντολή, έτσι όπως άλλωστε το ανέφεραν και κάποιοι συνάδελφοι που μίλησαν, ε, εντολή για ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την περίμετρο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η αρμοδιότητά μας είναι εγκάρσια, ε, όπως ε, μας εξήγησε άλλωστε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θυμάμαι ότι παλιότερα είχε υπάρξει και κάποια μελέτη η οποία αποτέλεσε την βάση για την ομοθεσία για τα δέσποτα ε, ζώα στην Ιταλία που κατεδείκνει ακριβώς την επίγουσα κατάσταση καταγράφοντας επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο που ε, τα δέσποτα ζώα μπορούν να έχουν όσον αφορά την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια, ακόμα και την οδική ασφάλεια. Ε, και μπορώ να συνεχίσω αναφέροντας και άλλα στοιχεία. Νομίζω ότι υπάρχει μία σειρά στοιχείων ανατομέα που μας δίνουν την υποχρέωση να προχωρήσουμε με τις αναφορές αυτές, να ζητήσουμε περαιτέρω στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως ε, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό και στους συντονιστές, ε, ίσως να ζητήσουμε και ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα το δούμε αυτό, ε, που θα βασιστεί αυτό το ψήφισμα στις πολλαπλές καταγγελίες που έχουμε από πλευράς των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, να σας ανακοινώσω ότι έχουμε ε, γνώση ότι θα φτάσουν και άλλες, πληθώρα μάλιστα, αναφορών με το ίδιο θέμα. Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως σκόπιμο θα ήταν να ζητήσουμε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε ε, να καταγραφεί ε, η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης χωρίς βεβαίως να ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες που έχουν τα κράτη-μέλη, τις εθνικές αρμοδιότητες. Θα δούμε, θα δούμε με τι εντολή θα συνεχίσουμε. Θα το αποφασίσουμε αυτό στη συνεδρίαση των συντονιστών. Πάντως, οπωσδήποτε, σκόπιμο είναι να κρατήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορές και να συνεχίσουμε μια πολιτικού χαρακτήρα πρωτοβουλία. Να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους αναφερόμενους ε, που μίλησαν, ήταν παρόντες. Ε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, και να ολοκληρώσουμε εδώ την συνάντηση της Επιτροπής μας. Ε, τρία λεπτά διάλειμμα και μετά θα συνεχίσουμε με τους συντονιστές.